Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Βλέπετε ότι εκ δεξιών ε, έχει έρθει ο Πάνος και χαιρόμαστε ιδιαίτερος όλοι. Η Βίκη το είχε αναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα του χρειαζόταν μια εβδομάδα για να ανανύψει γιατί είχε ένα δυστύχημα. Ε, πάντως χαίρομαι που ανέκαμψε και θυμάμαι και τις, ε, την κάρτα με τις υπογραφές και το, τις ευχές που στείλατε. Πάντως, ε, ηθικό δίδαγμα είναι ότι όταν είναι κανείς αυτοκίνητο, προσοχή. Πρέπει να έχει τα μάτια του 14, γιατί μπορεί ακόμη και τα ίδιος και το σφάλμα βαρύνει τον άλλον οδηγό, Παρ' όλα αυτά μπορούμε και εμείς να την πατήσουμε όσο προσεκτικοί και είμαστε. Προσοχή λοιπόν στην οδήγηση για να αποφεύγουμε τα τροχιά. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Η Ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Όχι, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας Υπενθυμίσω ότι αναμεταδίδεται και απευθείας ε, η συνεδρίασή μας από το διαδίκτυο. Να σας ενημερώσω επίσης ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της 27 η Απριλίου του 2016 έχουν ε, διανεμηθεί και αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. Συμφωνείτε? Λαμπρά. Θα ξεκινήσουμε από την ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Ανδρέα Σουάμπ, που είναι και ο μόνος επιζήσας από την ομάδα των σκιωδών εισηγητών και εισηγητριών που ε, ασχολούνται με το κείμενο. Άρα κανένα δεν πρόκειται να το διαβοψεύσει, μια και όλοι οι υπόλοιποι απουσιάζουν. Μπορεί να μα ενημερώσει για τι τριμερεί διαλόγου ό,τι αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από την ε, γνωμοδότηση που είχαμε ζητήσει, ανέλαβα στη θητεία αυτή το καθήκον ε, της ε, εισηγήσης και έτσι λοιπόν διοργανώθηκαν 10 τρισμερείς διάλογοι και 10 συναντήσεις των σκιωδών. Ήταν πραγματικά χρονοβόρα τη δικασία. Δαπανίσαμε πολύ χρόνο στο χαρτοφυλάκι αυτό, στο θέμα αυτό. Χαιρόμαστε λοιπόν όλος ιδιαίτερος και νομίζω ότι μιλάω εξ όλων των σκιωδών εδώ στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε λοιπόν που με το Συμβουλίο και με την Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα στις 25 Μαΐου καταφέραμε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου να καταλήξουμε σε μια λύση. Η μετάβαση σε ό,τι αφορά τα ιατρικά προϊόντα και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία in vitro, η μετάβαση λοιπόν από την οδηγία σε κανονισμό, αγαπητέ Πρόεδρε, σημαίνει σημαντικές αλλαγές των όρων πλαίσιο των συνθήκων πλαίσιων σε ό,τι αφορά τα ιατροφαρμακευτικά συστήματα, τα υλικά που συνδέονται με τις τεχνολογίες αυτές στην Βήτρο. Και ως εκ τούτου δεν, είναι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δυσκολεύτηκαν σε πολλά σημεία και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Γιατί ξέρετε από τις διαπραγματεύσεις κύριε Ροσφόρου στην προηγούμενη θετία, ιδιαίτερος η δική σας ε, είχε τα προβλήματα με τα εμφυτεύματα στήθους και έτσι τεθήκαν οι βάσεις για τις ε, τροποποιήσεις αυτές και τότε λοιπόν είπαμε με σαφήνεια ότι οι παραβιάσεις του νόμου δεν μπορούν να προκαλούν καινούριου ε, νόμους. Αλλά η παραγωγή τέτοιων προϊόντων θα πρέπει ποινικά να διώκονται, οι οποίοι δηλαδή ε, σκόπιμα και θελημένα παραβιάσαν την εμφιστάμενη νομοθεσία. Η βελτίωση ωστόσο των ε, μηχανισμών παρακολούθησης των εθνικών από τις εθνικές υπηρεσίες θα μπορούσε να βοηθήσει προκειμένου παραγωγή που ε, θέτουν στο εμπόριο επικίνδυνα προϊόντα να μπορούν να περιοριστούν. Και έτσι νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι είναι κάτι που καταφέραμε σε θέματα παρακολούθησης αγοράς στον, θέμα, στον τομέα των ιατρικών προϊόντων να το βελτιώσουμε και έτσι λοιπόν να γίνεται καλύτερη εποπτεία της παραγωγής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υψηλή επικοινωνιότητας προϊόντων. Αλλά αυτές οι βελτιώσεις, το τονίζω αυτό, μπορούν να επιδευτούν πραγματικά μόνο αν υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που προβλέπει ο Ευρωπαίος νομοθέτης. Και αυτό αφορά και την ενίσχυση των υφιστάμενων αρχών, γιατί αυτές θα κληθούν να αποδείξουν ότι έχουν δυνατότητα πραγματική εποπτείας και παρακολούθηση σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά. Δεν θα είναι όλα τα, προϊ... τα αρμόδια για την παρακολούθηση για τον έλεγχο των ιατρικών προϊόντων. Και ελπίζω λοιπόν να τεθούν σε μια προτεραιότητα για την κάθε χώρα και να υπάρξει συνεργασία. Και έτσι λοιπόν κάθε χώρα να έχει τον τομέα εξειδίκευσή του και έτσι στην τελική ανάλυση να υπάρχει όντω η προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τι 28 ξεχωριστέ εθνικέ αρχέ. Να υπάρχει παραπάνω προστιθέμενη αξία από ό,τι υπήρχε όταν, από όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Θα υπάρχουν επίση επιπρόσθετοι έλεγχοι για τα προϊόντα υψηλή επικίνδυνοτητα γιατί επικρίθηκε αυτό εν μέρη, αλλά σε κάποιους βασικούς τομείς, σε πραγματικά επικίνδυνων προϊόντων ή πολύ παρεμβατικών προϊόντων, στο μέλλον θα υπάρχουν πιο πολύ έλεγχοι. Μια προκαταβολική αδειοδότηση, μια προαδειοδότηση, προέγκριση δεν επιτρέφθηκε όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχει και πλέον ε, το ευρωπαϊκό σύστημα αδειοδότησης ε. εμφυτευμάτων. και για όλα τα ιατρικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν στα κράτη-μέλη καταφέραμε να βρούμε μία συμφωνία, ένα συμβιβασμό. Δεν είμαστε 100% ικανοποιημένοι, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρεί ότι ένας αρνητικός κατάλογος, ο οποίος δεν θα μπορεί να ανοίξει στην συνέχεια, σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πάντα θα έχει μια χρονική καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη νέων προϊόντων στο κατάλογο αυτό και αυτό ενδεχομένως να κατηγορηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καθυστερεί στην αντιδράσή της. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν διστακτική για την αποδοχή ενός τέτοιου αρνητικού καταλόγου. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει, από την άλλη δεν θέλει να παρακολουθήσει και την, ε, το συμβιβασμό μεταξύ των δύο νομοθετών, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και αυτός ο τρομερής διάλογος ε, θεωρώ ότι τελικά θα καταλήξει σε ένα συμβιβασμό ο οποίος θα πονέσει και τις τρεις πλευρές. Αλλά αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιβαρυνθεί υπερβολικά η κοινοτομική αυτή βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος εκεί που χρειάζεται στους ε, τομείς υψηλή επικινδυνότητας για του ασθενεί. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θεωρώ λοιπόν ότι επικοδομητική ήταν η στάση του Κοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν σε τελική ανάλυση και οι συνάδελφοι να μπορέσουν να εγκρίνουν το συμβασμό αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σουάπ. Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και δεν μπορούμε ε, έτσι επιπόλαια να προσεγγίζουμε κείμενα ή απροετοίμαστοι. Και χαίρομαι που αργά αλλά σταθερά καταλήγουμε σε συμβαστικέ τροπολογίες και συμφωνίες, παρόλο που δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικέ ε, απόλυτα για όλους, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την εποπτεία μετά σε ό,τι φορά την εφαρμογή των κανόνων. Υπάρχουν σχόλια για την ενημέρωση που μα έκανε ο κ. Σβάμπ. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πάντως θερμά τον κύριο Σφάπ για το έργο του που δεν έχει ακόμη διεκπαιρεωθεί, αλλά προχωρεί με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο που αφορά την έκθεση για την έγκριση και υποπτήρια της αγοράς ε, για τα οχήματα ε, μηχανοκίνητα και τα τους του, ε, τα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και τι χωριστέ τεχνικέ μονάδε του. Ο κύριο Ντάλτον είναι ο εισηγητή μα. Και μάλιστα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, με ενδιαφερομένου. Γι' αυτό και έχουμε ένα πάνελ ε, με καλεσμένους που θα λάβουν διαδοχικά το λόγο και θα σας τους παρουσιάσω στον έναν ανά με τη σειρά. Ο κύριος Ντάλτον όμως θα μας κάνει πρώτα μία εισαγωγή πριν περάσουμε στην ακρόαση με τους ενδιαφερομένους. Ο κύριος Ντάνιελ Ντάλτον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι καλό που επιτέλους γίνεται σωστή συζήτηση με τους ενδιαφερομένους. Δεν είχαμε πολύ χρόνο όσον αφορά αυτή την έκθεση και όπως μου είπαν και κάνα δύο άλλοι σκιώδεις πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε το θέμα. Είναι σημαντικό νομοθέτημα και είναι λίγο απογοητευτικό που είναι Δευτέρα πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, διότι δυστυχώ δεν είναι τόσοι παρόντε όσο θα έπρεπε. Επευθυνώ έκκληση προ τη γραμματεία, μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάπω το χρονισμό στο μέλλον. Πέραν αυτού, προσβλέπω στο να ακούσω τι θα πούν οι ενδιαφερόμενοι. Έγινε κάποια συζητήση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ακούσαμε την άποψη των άλλων ενδιαφερομένων. Θέλουμε να ακούσουμε τι θα πούνε. Θα προτιμούσα να του δώσω το λόγο και να πάρω το λόγο εγώ αφού πάρουν εκείνοι το λόγο και του ακούσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντάλτον. Δίκιο έχετε όσον αφορά τα δύο που είπατε. Πράγματι θα πρέπει το κείμενο να συζητείτε και αντιμετωπίζετε όταν είναι εδώ οι βουλευτέ. Δεν φταίνει η γραμματεία αν δεν έρχονται εδώ εγκαίρω οι βουλευτέ, ή όταν ξεκινούν οι συνεδριάσει τη επιτροπή. Θα δώσουμε το λόγο αμέσως στους ενδιαφερομένους σας ζητούμε, σας παρακαλούμε αν μπορείτε να περιοριστείτε σε ένα εξάλεπτο στις παρουσιάσεις σας. Ο κ. Άλμπερτ Κλός είναι πρώτος. Ε, από την Ένωση των κατασκευαστών ε, αμαξωμάτων ε, διαφόρων οχημάτων. Κύριε Κλώζ, έχετε το λόγο. Είναι εκτός μικροφώνου ο κ. Κλώζ, δυστυχώς δεν ακούμε. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ να μιλήσω στο Κοινοβούλιο. Είμαι ο Αλφατ Κλός, τεχνικός διευθυντής της ΙΑΕ, επιφορτισμένος για να συμμορφωνόμαστε με τον κανονισμό πλαίσιο. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι καλωσορίζουμε την πρόταση κανονισμού και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θέλουμε οι δυσκολίες του τρέχοντος συστήματος να διορθωθούν. Όμως, σημαντικό για μα είναι οι νέε προτάσεις να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά το κόστος και να μην αυξάνουν τη γραφειοκρατία. Συγγνώμη, ξέρετε είμαι λίγο ταραγμένος που μιλάω δημοσίω. Μα δίνεται η δυνατότητα μέσω τη να απλουστεύσουμε το παρόν σύστημα. Ταυτόχρονα μπορούμε να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά για την έγκριση των οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντοπίσαμε κάποια κρίσιμα σημεία, μεταξύ αυτών θέτω επί της οθόνης 2. Καταρχάς, το πενταετές όριο για την ισχύ των πιστοποιητικών. Αυτό μπορεί να γίνει τεράστιο πρόβλημα για την βιομηχανία. Διότι για τις αρχές και τους κατασκευαστές διότι ε, ε, μια τέτοια έγκριση τύπου δεν αφορά μόνο το σύστημα όλο του οχήματο, αλλά έχουν περίπου 400 συστήματα σε ένα μεγάλο φορτηγό. Κάθε όχημα έχει διαφορετικά συστήματα. Και να εγκρίνουμε όλα τα συστήματα ξεχωριστά κάθε πέντε χρόνια δεν είναι τόσο εύκολο. Δεύτερον, η χρηματοδότηση της αγοράς εγκρίσεων τύπου και τη εποπτείας αυτή μέσω ενός συνδυασμένου εθνικού τέλους εισφοράς. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν τόσες πολλές εγκρίσεις τύπου να κάνουν. Ένα-δύο οχήματα εγκρίνουν στη χώρα τους και εξακολουθούν να έχουν τεράστιο βάρος όμως για την εποπτεία της αγοράς. Η κατανομή του βάρους εποπτείας της αγοράς σε δύο εγκρίσεις τύπου το κόστος το κάνει απαγορευτικό για τις εγκρίσεις τύπου και οδηγεί στην προσπάθεια εξέβρεσης της φθηνότερης εγκρίσεως τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν και κάποια μέτρα προβλέπονται που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Όπως σε μη, μη κρίσιμες μη και μεγάλη γραφειοκρατία. Διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να επιληθούν διοικητικά. Λοιπόν, κλείνοντας, εμείς σαν ΑΣΕΑ θέλουμε να συμμετάσχουμε στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Θέλουμε να συζητήσουμε και να υποστηρίξουμε κάθε επικοδομητική πρόταση. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε προτάσεις για την πρόληψη της συνέχισης των υφισταμένων τύπων οχημάτων που θα οδηγούσε σε μία ε, μη εφαρμογή των απαιτήσεων. Επεξεργαζόμαστε προτάσεις για τη χρηματοδότηση της εποπτείας της αγοράς χωρίς να δημιουργούμε οικονομικές εξαρτήσεις που θα, δημιουργούν θα καταστρέφουν μάλλον τις ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Και τέλος, θέλουμε να συνεργαστούμε κρισίμων θεμάτων που θίγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κλώσ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρχαρτ Μίλλερ που είναι ε, από την ε, Διεθνή Επιτροπή ε, Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα που ασχολείται με την επιθεώρηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Σας δίνω το λόγο κύριε Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος ε, της ομάδας εμπειρογνωμόνων της, Επιτροπή της Επιτροπής για τη χορήγηση εγκρίσεων ε, στη ΣΥΤΑ, τη Διεθνή Επιτροπή Επιθεώρησης Μηχανοκίνητων Οχημάτων, θα θέλουμε να χαιρετήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία να έχουμε μια πιο επαγγελματική προσέγγιση αυτών των συστημάτων στο μέλλον. Θα σας παρουσιάσω συντομία κάποια σημεία. Καταρχήν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ανάγκη μια ομοιόμορφη ε, μετάθεση στην εθνική νομοθεσία των διαφόρων νομοθετικών διατάξεων. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε ήδη το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, που ρυθμίζει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο τις σχέσεις ε, μεταξύ κατασκευαστών και καταναλωτών. Δεν είναι σκόπιμο λοιπόν στο μέλλον ε, οι τεχνικές υπηρεσίες να ε, αποκτούν εντολή και για την ε, τυποποίηση, τη χορήγηση έγκρισης. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, τα διάφορα, με τις διάφορες δοκιμές. Τα κατασκευαστικά στοιχεία είναι χιλιάδες μερικές φορές και τα ανταναλλακτικά. Επίσης έχουμε διαφορετικές ε, δομές ε, τιμών μεταξύ των κρατών μελών. Και στην έμπρακτη εφαρμογή υπάρχει πολλές φορές πρόβλημα. Και μεγάλη γραφειοκρατία και διατυπώσει, ε, αν θεσπίσουμε συγκεκριμένε και μεμονωμένε διαρθρώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια εναρμόνιση των απαιτήσεων, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε διάφορου κανόνε σχετικά μειόμορφους, που μπορούν να είναι πιο λεπτομεριακοί και δελεχείς και επίσης έχουμε και ένα checklist ε, με, τον ακριβή, με την ακριβή περιγραφή των ελάχιστων προδιαγραφών για τις διάφορες τεχνικές υπηρεσίες. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και θα ενισχύσουμε την, τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία τους. Επίσης θέλουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων ε, υπευθύνων. Έχουμε τις αρχές αναγνώρισης, τεχνικές υπηρεσίες, έχουμε τους ε, κατασκευαστές ε, αυτοκινήτων. Τρεις κατηγορίες τελεστών που θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες μεταξύ τους, ώστε να μην έχουμε μια κατάσταση σαν τη σημερινή, όπου μια αρχή να μπορεί να εξασφαλίζει και την τεχνική, τις τεχνικές υπηρεσίες και τον τεχνικό έλεγχο. Επίσης θέλουμε και μια γενική υποπτία της αγοράς σε όλη τη διάρκεια ζωή, από την αρχή δηλαδή μέχρι την έγκριση. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθεί ο τομέα εφαρμογή και να υπάρχει και το conformity of production, ε, η συμβατότητα του προϊόντο και το in-service conformity. Αυτό να διεξαγαγείται από τρίτου ανεξάρτητε υπηρεσίε. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η δεσμευτική διεξαγωγή ελέγχου των ε, οχημάτων σε ό,τι αφορά τα αυτοματοποιημένα, στην, τα οχήματα αυτοματοποιημένης μετακίνησης. Και εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε την ε, κατάσταση του λογισμικού για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ε, παρεμβάσεις ε, και χειραγωγήσεις. Και θεωρούμε ότι σημαντικό είναι να δούμε τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων και εδώ πέρα θα γίνει ε, σύνδεση μεταξύ των έλεγχο, των, με το ελέγχου τύπου και την ε, σωστή εξαγωγή ελέγχου στα τακτικά χρονικά διαστήματα. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε εξ αρχής από την έγκριση του τύπου σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές ελέγχου, οι οποίες θα πρέπει να οριστούν για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να οριστεί είναι ότι τέτοια έλεγχοι οι οποίοι γίνονται κάθε εκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνονται χωρίς αποσυναρμολόγηση των οχημάτων. Ιδάλλως είναι τεράστιο το κόστος για τον καταναλωτή. Δεν μπορεί να καλυφθεί. Ένα τελευταίο ζήτημα. Ένα φόρουμ συντονισμού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μεταξύ όλων των φορέων όχι μόνο των εποπτικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών θα γίνεται τακτική ανταλλαγή πληροφοριών. Και ότι υποπίπτει στην ε, προσοχή του καθενός θα επισημαίνεται σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αμφιβολία για τη σωστή λειτουργία Άρα, συνοψίζοντα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν τεχνικά πρότυπα αναρμονισμένα και μάλιστα σε πιο υψηλό επίπεδο αναρμόνιση. πρόσβαση στο λογισμικό και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και η ενσωμάτωση, η ενοποίηση μάλλον των ε, ελέγχων στον περιοδικό έλεγχο οχημάτων. Σας ευχαριστώ. Ναι, διαπιστώνουμε και από την επικαιρότητα τι στρατηγική σημασία έχει αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε με τους επαγγελματίες στον τομέα του αυτοκινήτου. Το ρόλο έχει ο κύριος Ιάκομπ Μπάνξκαρ, που είναι ο Διευθυντής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων. Φαντάζομαι εδώ καλύπτουμε το σύνολο του κλάδου, όχι μόνο τις τεχνικές πτυχές. Έχετε το λόγο, κύριε Μπάνξκαρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να παρίσταμε σήμερα. Είμαι υπεύθυνο στο φορέ μας για δραστηριότητες κινητικότητας στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και σήμερα μιλώ εκ μέρους των 75 Ευρωπαίων ε, συλλόγων ε, κίνησης που εκπροσωπούν περίπου 75 εκατομμύρια ε, μέλη. Έχουν δικαίωμα καταναλωτέ να έχουν ακριβεί πληροφορίε για τα προϊόντα που αγοράζουν και για την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων και αυτό δεν ισχύει πάντα. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μα και η κινητικότητα, ο τομέα κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό και πώς αυτή η αναθεώρηση μπας συμβάλλει σε αυτό, μπορεί να βελτιώσει τα συστήματα εγκρίσεων τύπου και μπορεί να εισάγει ε, μέτρα για την επαπτή υποπτία της αγοράς. Το σύστημα εγκρίσεως τύπου καθορίζει κάποιες κοινέ προϋποθέσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον, εξασφαλίζει αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου και ελεύθερη διακίνηση των α, ε, οχημάτων. Το παρόν σύστημα εγκρίσεως τύπου υποστήριξε την αρχή της ενιαίας αγοράς, Βελτίωσε την οδική ασφάλεια, όμως απέτυχε σε τομείς όπως τα ωφέλη για το περιβάλλον. Η εμπειρία τι καταδεικνύει, ότι η άμεση οικονομική σχέση μεταξύ των κατασκευαστών και των συστήματων εγκρίσεως τύπου και τεχνικού ελέγχου στρεβλώνει την αγορά. Χρειάζεται ξεχωριστή δομή ε, εισφορών να μην επηρεάζουν οι κατασκευαστέ τις άλλε αρχέ εγκρίσεων τύπου και από τη αγορά, όμω η πρόταση χρειάζεται να ρυθμίσει λεπτομέρειε για να μειωθεί το κόστο και να είναι αποτελεσματικότερο το σύστημα. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτρέπει και στα κρατημέρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλουν κυρώσει και διοικητικά πρόστιμα είναι ένα καλό βήμα πρόοδου, Σαφεί ευθύνε και σαφή βήματα να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση μπορεί να προστατεύσει τον καταναλωτή, ώστε ο καταναλωτή να μην λαμβάνει ανακριβεί πληροφορίε για τα προϊόντα που αγοράζει. Η πρόσβαση στα στοιχεία για συμμόρφωση, για επαλήθευση συμμόρφωση και πρόσβαση στο λογισμικό χυμάτων είναι άλλο σημαντικό βήμα. Οι πληροφορίε θα πρέπει να διατίθεται σε επιλέξιμου ε, ελεγκτικού φορεί. Θα πρέπει να γίνονται δοκιμέ και έτσι να εξασφαλίζεται ότι έχουμε επαρκείς αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για τους καταναλωτές. Τώρα, σαν αφορά την εποπτεία της αγοράς, η ιστορία έχει δείξει ότι χρειάζεται να γίνονται μεγαλύτερες, περισσότερες επαληθεύσεις από τη στιγμή που διτίθεται τα οχήματα στην αγορά. Εμείς στην FIA μαζί με τα μέλη μας συμμετέχουμε ενεργά στις δοκιμές για θέματα ασφαλείας και περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων όταν φτάσουν στις αντιπροσωπείες. Θα θέλαμε να δούμε επαρκείς φυσικές δοκιμές που θα γίνονται και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πληροφορίε που απαιτούνται για τις δοκιμές θα πρέπει να διατίθεται σε ανεξάρτητα τρίτα μέρη, ούτω ώστε να γίνεται δοκιμή ανεξάρτητη ατελώ και άμεσα. Οργανισμοί ανεξάρτητα θα πρέπει να κάνουν δοκιμές τακτικά και να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα άμεσα στο σωστό φορέα επιβολής και συμμόρφωση. Οι καταναλωτέ θα πρέπει να έχουν διαφανεί πληροφορίε στη θέση του από τι δραστηριότητε για την εποπτεία τη αγορά. Κάτι τελικό που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα είναι το εξή ότι τα οχήματα πολύ γρήγορα μπαίνουν σε ένα νέο τομέα με αυξανόμενο αυτοματισμό και διασυνδυσιμότητα και η έγκριση τύπου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχουν ισότιμες συνθήκες για τις πληροφορίες, για τη συντήρηση και επισκευές και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την εποχή που έρχεται. Λοιπόν, Έχουμε νέε δυνατέ επικοινωνίε για τα οχήματα. Χρειαζόμαστε νέο πλαίσιο για επιλογή για του καταναλωτέ, για τον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και για την προστασία των δεδομένων. Ενθαρρύνουμε θερμά το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί του Ευρωπαίου καταναλωτέ να εξασφαλίσει ότι επαρκή μέτρα συμμορφώσεω θα θεσπίζονται και θα εφαρμόζονται ταχύτερον δυνατόν, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Μπάνσκαρτ. Δύο ακόμη καλεσμένοι μας έχουν απομείνει, δύο γυναίκες μάλιστα. Θα δώσω πρώτο λόγο στην κυρία Σίλβια Γκάτζετ, που είναι η εκπρόσωπος της ΑΦΚΑΡ, που είναι η Συμμαχία για την Ελευθερία της Επισκευής Αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ο τίτλο αυτής της οργάνωσης ε, και μας δίνει μια ιδέα, μας προειδάζει για το τι θα ακολουθήσει. Περιμένουμε και τι δικέ προτάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη θέση μου. Ε, μία από τις πολλές πτυχές ε, της ε, έγκρισης τύπου για το αυτοκίνητα αφορά και τις πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση του αυτοκινήτου, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της Ένωση μας. Είμαστε η Συμμαχία για την Ελευθερία της Επισκευής Αυτοκινήτου. Ήδη δημιουργηθήκαμε από το 1997 και έχουμε μια ευρία γάμα ενδιαφερομένων από τη ΦΙΑ, τους αυτοκινητοβιομηχανίες και την αγορά ε, κατόπιν από την, την Αιτζία, τη ΦΙΤΖΙΕΦΑ, ΑΤΦΑ, καθώς και ΑΤΦΑ, καθώς και τη ΣΕΚΡΑ, που είναι οι ανεξάρτητοι επισκευαστές. Θέλουμε ε, ένα θεμητό ανταγωνισμό για τα αντανακλαστικά αυτοκινήτων, για τους ε, τεχνικούς ελέγχους, ε, τις υπηρεσίες και τις επισκευές και, και δίκαιη πρόσβαση. Γιατί σε αυτό το τομέα της μεταπόλησης απασχολούνται 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι και είναι κυρίως μικρομεσαίες αυτές οι επιχειρήσεις που αποτελούν τμήμα της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας και μάλιστα ε, προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες συντήρησης και επισκευές ε, στους 284 εκατομμύρια καταναλωτές και χρήστες αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ο σχετικό κανονισμό για τι εγκρίσει τύπου και την επίτευξη τη αγορά ουσιαστικά ενοποιεί τι προηγούμενε διατάξει για τι πληροφορίε που δίνονται για τη συντήρηση, το RMI, για, από τον κανονισμό Euro 5 για τα επιβατικά και το Euro 6 για τα επαγγελματικά οχήματα. Η πρώτη μου παρατήρηση πάντως αφορά κάποιες παραλήψεις ε, του κανονισμού. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά το OBD, αυτό το σύστημα, το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης ε, προβλημάτων, που θα πρέπει να δίνει πληροφορίες και γι' αυτό αυτή η στάνταρ σύνδεση θα πρέπει να επανέλθει. Επίση, αναπρογραμματισμός, των προδιαγραφέων για τα επιβατικά αυτοκίνητα θα πρέπει να τη χάνει ε, τακτικής ενημέρωσης. Επίσης, ε, για τα επαγγελματικά φορτηγά, βαρέα επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να ε, επαναντάξουμε αυτές τις διατάξεις και άλλες που λείπουν σε αυτή τη διαδικασία που υπάγεται στη συναπόφαση. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη σχετική διαφάνεια. Και εκτός του, της επαναφοράς των παραλήψεων θα πρέπει να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις που είναι απολύτως απαραίτητες ώστε το σύστημα για την πρόσβαση στην τεχνική ε, ενημέρωση να γίνει πιο στιβαρό και εύχριστο σε πρακτικό επίπεδο. Είναι ήδη παλιά η υφιστάμενη νομοθεσία, είναι δεκαετής και θα πρέπει να τύχει κάποιες επικαιροποίησεις ε, για να ανταποκριθεί στις νέες ε, καταστάσεις. Η έκθεση Ρικαρντό για την λειτουργία του συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2014. Εκεί εντοπίζονται κάποιες διαφορετικές ε, ανεπάρκειες και προβλήματα εφαρμογής. Φάνηκε για παράδειγμα ότι οι επισκευαστέ, αλλά και η αλυσίδα ε, παροχής υπηρεσιών ε, μετά την πώληση προσκρούει σε εμπόδια από την αυτοκινητομηχανία που δεν εξασφαλεί πρόσβαση ε, σε τέτοιες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν απολογισμό 160 προβλημάτων με συστάσεις για το πώς θα βελτιωθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός για την έκρηση τύπου. Μάλιστα, τα μέτρα που ακολούθησαν τη έκθεση Ρικάρντο δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί επισήμω στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ώστε να κλείσουν τα παραθυράκια που οδήγησαν σε μία αναποτελεσματικότητα στο, σύστημα πρόσβασης, στο ισχύο σύστημα πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, για να εξασφαλίσουμε διαθεσιμότητα ε, ενός ε, διαγνωστικού συστήματος ε, για πολλές μάρκες θα πρέπει να έχω μια έγκριση του interface του του, αυτο, του οχήματος. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ανεξάρτητα εργαλεία ελέγχου που θα πρέπει να υπάγονται σε στάνταρ πρωτόκολλα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ομοιομορφία. Με βάση την έκθεση Ρικάρντο, μερικοί ε, κατασκευαστές δεν απαντούν στις ε, αιτήσει έγκρισης. Μάλιστα έχουν αποτρεπτικά τέλη ή δεν ε, ε, χορηγούν πληροφορίες για το περιβάλλον του ελέγχου. Θα πρέπει η αυτοκινητοβιομηχανία μέσα σε ένα εξάμεινο να χορηγήσουν αυτό το test environment, κάτι που δεν κάνουν. Επίσης, ο ορισμός ε, για την συντήρηση είναι το 2006. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί για να περιλάβει και το κατασκευαστή ως νέο τελεστή της αλυσίδας ανεφοδιασμού. Και οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται με τη μορφή που να επιτρέπει την ηλεκτρονική τους επεξεργασία. Γιατί πολλές ιστοσελίδες ε, δεν είναι καθόλου φιλικές ε, για το χρήστη και για πολλούς τελεστές της αλυσίδας εφοδιασμού. Κάτι που απάδει από τις ε, προθέσεις του κανονισμού. Επίσης, καλούμε το Κοινοβούλιο ε, να ενισχύσει τα συστήματα έγκρισης και εφαρμογής και να ε, απλουστευτεί η διαδικασία καταγγελίας και επιβολής αιτιάσεων. Γιατί η παρούσα διαδικασία είναι παχθής για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Φανταστείτε τι Πώς είναι δυνατόν ένας Ολλανδός φορέας να επεξεργαστεί ε, μια καταγγελία που γίνεται από, μια βουλγαρική, από ένα βούλγαρο καταναλωτή για ε, ένα αυτοκίνητο που έτυχε έγκριση τύπου στη Βουλγαρία. Θα πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε αυτό το κενά και να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών, αυτών που εξασφαλίζουν τον έλεγχο και αυτών που έδωσαν την έγκριση τύπου, ώστε να γίνεται δυνατή διερεύνηση ε, υποθέσεων προβληματικών. Η ΑΦΚΑΡ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προασπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, και τους 285 οδηγούς αυτοκινήτων, κυρίως για τη μεταπολιτική περίοδο και για την ελεύθερη επιλογή του επισκευαστή. Θα πρέπει επίση να διορθωθούν οι αδυναμίε του υπάρχοντο συστήματο και να εξασφαλιστούν, να διατηρηθούν οι συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού. Επίση, ε, δεν θα πρέπει αυτό να, να, να το μπερδέψουμε με το σύστημα ψηφιακή πρόσβαση. Γιατί ε, χρειαζόμαστε μια ε, διασυνδέσιμη τηλεματική πλατφόρμα και αυτό είναι το αντικείμενο μια ε, μελέτη που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Ιούνιο. Πιστεύουμε ότι έτσι θα δημιουργηθούν οι βάσει για μια πιο ε, περιεκτική αναθεώρηση του κανονισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και ανάγκε τη ψηφιακή εποχή. Βέβαια θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ε, σημερινής εποχής, αναλογική και των εμποδίων που υπάρχουν. Στο κυρία μου ήταν πάρα πολύ σαφής η παρουσίασή σας. Τέλος για να ολοκληρώσουμε αυτό είναι επισκόπηση. Η κυρία Σίλβια Μορέρ έχει το λόγο. Εκπροσωπεί το ΜΠΕΚ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προασπίσεως των Δικαιωμάτων Καταναλωτού και θέλει να μιλήσει για το θέμα της βιωσιμότητας ασφάλειας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΙΜΚΟ που κάλεσε την ΠΙΟΚ να συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων. Από πλευράς καταναλωτών η ΜΠΕΚ εκπροσωπεί 42 ανεξάρτητους εθνικούς φορείς καταναλωτών από 31 ευρωπαϊκές ε, χώρες και αυτό που μας ενώνει βασικά είναι ότι τα μέλη μας, τα μέλη της ΜΠΕΚ θέλουν πραγματική δράση για την εποπτεία της αγοράς των αυτοκινήτων και τις εγκρίσεις τύπου αυτοκινήτων στο μέλλον, πώς θα κινηθούμε όχι μόνο με το σκάνδαλο για τα διζελοκίνητα, βρήκαμε και άλλα πολλά κενά και έχουμε σοβαρές ανησυχίες ότι τα δικαιώματα και συμφέροντα των καταναλωτών δεν γίνονται σεβαστά από κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, αν οι εκπομπέ είναι πολύ ψηλέ, αλλά και πρόβλημα για το πορτοφόλι του καταναλωτή, αν τελικά δεν ανταποκρίνεται η κατανάλωση του αυτοκινήτου στι προσδοκίε του αγοραστού. Γι' αυτό επίση η Άλτρο Κοσούμου, Ιταλικό μα μέλο, ξεκίνησε προσφυγή στην Ιταλία το 2015 για να βοηθήσει του ιδιοκτήτε αυτοκινήτων δύο μοντέλων να πάρουν πίσω τα χρήματά του. Διότι θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα οικονομικό, συν τη άλλη. Προφανώ, όπω ακούσαμε, το Κοινοβούλιο λέει ότι χρειάζεται χρόνο για συζητήσει. Το κατανοούμε. Είναι σημαντική σοβαρή συζήτηση και ο κατάλληλος χρόνος για τη λήψη αποφάσεων. Όμως, απευθύνω μια έκκληση. Πρέπει να προχωρήσουμε, χρειάζεται. Πρέπει να προσεχθεί το θέμα, όλος ιδιαίτερος. Διότι για την ώρα κάποιοι πολίτες έχουν αμφιβολίες όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που δίνει η Ευρώπη για τον απλό πολίτη. Αν εδώ πετύχουμε αποτελέσματα, μπορούμε να έχουμε ορατότητα όσον αφορά την Ευρώπη. Ότι μπορεί η Ευρώπη να καλύψει κάποια κενά. Αυτό μπορούμε να δείξουμε. Να πω ότι πριν την ανταλλαγή των απόψεων έχουμε εκδώσει ένα έγγραφο με τις συστάσεις μας, εκφράζει τη θέση μας. Να συνοψίσω κάνα δύο σημεία δικά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε έκανε πολύ καλή πρόταση. Μεγάλο βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Όμως για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αυτοκινητοβιομηχανία, καλούμε το Ευρωκοινοβούλιο να ε, επιβάλλει κάποιες απαιτήσει. Θα πρέπει να γίνονται τυχαίες δειγματοληπτικές δοκιμές στα αυτοκίνητα, να δούμε αν υπάρχει συμμόρφωση όταν κινούνται τα οχήματα στους δρόμους, και θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερη σχέση μεταξύ κατασκευαστών εθνικών αρχών και φορέων δοκιμών, όπως ανέφεραν και κάποιοι προλελήσαντες. Πιστεύουμε ότι μόνο συνδυασμός ελέγχου των νέων μοντέλων αυτοκινήτων και δοκιμών των οχημάτων όταν κινούνται στον δρόμο, αυτά θα εξασφαλίσουν ότι θα έχει εμπιστοσύνη ο καταναλωτής στο αυτοκίνητο που αγοράζει και το νομικό κείμενο τελικά πρέπει να καθορίζει ελάχιστο αριθμό οχημάτων που θα πρέπει να επαναξεταστούν μετά την αγορά τους από τους καταναλωτές. Τι παρατηρήσαμε, ότι υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά το παρόν σύστημα εγκρίσεων τύπου και αυτή αναθεώρηση σημαντική ευκαιρία να διορθωθούν όλα αυτά. Όλοι οι ιδιωτικέ τεχνικέ υπηρεσίε που ελέγχουν τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εξάρτητοι φορεί από την βιομηχανία και από του παρόχου και του πολιτέ ανταλλακτικών. Και οι δοκιμέ θα πρέπει να γίνονται ε, σε ανεξάρτητα εργαστήρια. Έχουμε και άλλη μια σύσταση. Ότι οι ιδιωτικέ τεχνικέ υπηρεσίε δεν θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές από τους κατασκευαστές και οι κατασκευαστές δεν θα πρέπει να επιλέγουν τη τεχνική υπηρεσία. Κάποιος φορέας Ευρωπαϊκής Ενώσεως ιδιωδός ή κάποιος άλλος φορέας θα πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι μια σύσταση που κάπως διαφέρει από τους προηγούμενους ομιλητές σαν τοποθέτηση. Ένα σημαντικότατο θέμα για μας χρειάζονται πάρα πολύ καλές διατάξεις για τις πινές, για τις κυρώσεις. Θα πρέπει να καλύπτεται κάθε μορφή μη συμμόρφωσης. Ακόμα και όταν η κατανάλωση των καυσίμων, η κατανάλωση δεν ευθυγραμμίζεται με τα επίσημα στοιχεία των δοκιμών. Πρέπει επίσης να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι και η χρήση συσκευών που ξεγελούν τις δοκιμές είναι κάτι παράνομο. Όσο έχει το κείμενο τώρα δεν το ξεκαθαρίζει. Πρέπει να ενισχυθεί η διατύπωση. Είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να επικρατεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εγκρίσεων τύπου. Πρέπει να εξασφαλίζουμε μεγαλύτερο έλεγχο και λογοδοσία από πλευρά αρχών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, να ελέγχονται οι τεχνικέ υπηρεσίε και οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων. Έχουμε πρόβλημα να έχουμε πρόσβαση στι πληροφορίε τώρα και ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Όταν εξετάζουμε ζελοκίνητα το σκάνδαλο στα ζελοκίνητα Καμιά φορά δεν ξεκάθαρο γιατί μια ανάκληση είναι ε, υποχρεωτική σε μια χώρα και σε άλλη χώρα δεν είναι. Θα πρέπει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα νέο σύστημα και να υπάρχει μια ομοιόμορφη απάντηση στις μη συμμορφώσεις. Στη δημόσια συζήτηση αναφέρεται συχνά ότι τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Επίσης, και οι οδηγοί υποφέρουν περισσότερο όταν είναι πολύ ψηλές οι εκπομπές, διότι τα αέρια των εξατμίσεων εισέρχονται και στο όχημα και τον απνέουν οι χρήστες του αυτοκινήτου. Οπότε είναι προς όφελος των καταναλωτών να μην γίνεται αυτό. Πρέπει να πω ότι καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα φόρουμ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών θα ήταν καλό να προβλέπετε ρητά ότι οι οργανώσεις των καταναλωτών θα μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, διότι τα μέλη μας εξετάζουν αυτοκίνητα σε εργαστήρια, έχουν εντοπίσει περιπτώσεις μη συμμορφώς κατά το παρελθόν που θα θέλαμε τις περιπτώσεις αυτές να μπορούμε να σκηνοποιούμε σε ένα τέτοιο βήμα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ακούσαμε λοιπόν τους πέντε προσκεκλημένους που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους φορείς, θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Ο κ. Στέφανεκ ήδη είναι έτοιμος να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω, όχι. Α. Ο Κρυστάλ Σάντελμος, Σκιώδης των Σελιστών, έχει παρε... κάποιες παρατηρήσεις. Θέλει Κριστάλ να πάρει το λόγο. Άμα δεν θέλει, δεν είναι σοβαρό. Θέλετε. Τι σκιώδης έχω απέναντί μου. Ορίστε, σα δώσω, σας δώσω το λόγο. ίσως ο κ. Στέφανεκ μπορεί να μιλήσει μετά. Κριστέλ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο στην παρουσιά φάση και νομίζω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και θα εμαθύνουμε ενδεχομένω. Πρόκειται για κάποια εισαγωγικά σχόλια και μόνο εμείς ως σοσιαλδημοκράτες πιστεύουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια καλή βάση μια καλή βάση για την βελτίωση των συστημάτων έκρησης τύπου. Και αυτό αποτελεί μια πραγματική ανάγκη, μια πραγματική έλλειψη. Θα πρέπει να υπάρξει αυτή η βελτίωση, θα πρέπει να φροντίσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Να μπορούν να βασίζονται στο σύστημα παραγωγής αυτοκινήτων και προκειμένου να υπάρχει ασφαλώς και δίκαιος ανταγωνισμός για τους αυτοκινητοπαραγωγούς. Ωστόσο, είναι παράλληλα εξίσου σημαντικό στο μέλλον να ερευνήσουμε το τι γίνεται με τα δεδομένα στα οχήματα, στα αυτοκίνητα, η πρόσβαση στα δεδομένα αυτή στα δεδομένα αυτά, ε, η ασφάλεια των δεδομένων αυτών και όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε λοιπόν. Και ασφαλώς και το θέμα των κυρώσεων. Μας απασχολεί ιδιαίτερα. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον το εφιστάμενο σύστημα είναι το πλέον ευνοϊκό, το πλέον δεδειγμένο. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον κάθε κρίκος της αλυσίδας γνωρίζει επακριβώ το τι θα πρέπει να κάνει και το ποια είναι τα καθήκοντά του. Σε ό,τι αφορά την έγκριση του τύπου, σε ό,τι αφορά την υπηρεσία περιβάλλοντος, ε, το ΔΕΚ, να ξέρουν ε, Όλοι λοιπόν ε, ποιο είναι ο τους προκειμένου ε, να αποφύγουμε και ενδεχόμενο μελλοντικό τέτοιο σκάνδαλο. Επίση, θα κληθούμε να ορίσουμε το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Τι είδου στρατηγικέ ε, ε παρέμβαση και χειραγώγηση επιτρέπονται και ποιε όχι. Δύο λόγια τώρα για το χρονικό τη χρονική διάσταση σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Κατανοώ ότι είναι πραγματικά επιγόντω να αναθεωρήσουμε το σύστημα έγκρισης τύπου. Αυτό το οφείλουμε και στον καταναλωτή και στον πολίτη γενικότερα. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε όλα αυτά να συμβούν σωστά και ορθά. Υπήρξαν λοιπόν τα σκάνδαλα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε το σωστό χρόνο στην έρευνα του τι πήγε λάθος. Πώς είναι δυνατόν να μην ανακαλύφθηκαν τα σκάνδαλα αυτά καν στην Ευρώπη, να καταλήξουμε τελικά να τα ανακαλύψουν αυτά οι Αμερικανοί. Είναι ερωτήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Βιαζόμαστε μεν, αλλά θα πρέπει να αφιερώσουμε το χρόνο που χρειάζεται. Η σωστή και εις βάθος έρευνα των ζητημάτων αυτών. Χαίρομαι επίσης και προσβλέπω στην καλή συνεργασία και είμαι βέβαιη ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα εξαιρετικό σύστημα και για τους καταναλωτές αλλά και για τους παραγωγούς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κυρία Σάλντε Μόζα ότι οι ερωτήσεις που θίξατε αναλύονται στην Διερευνητική Επιτροπή εμείς ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο με τα τζελοκίνητα της Volkswagen. Δεν ξέρω αν θέλει και ο κύριος Εκ α, να λάβει το λόγο. Όχι, ο Ανδρέας Σαπ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το γεγονός ότι μας παρουσιάσατε σήμερα με πολύ επακριβή τρόπο ποια είναι η άποψη των εμπλεκομένων φορέων και θα συμφωνήσουμε με την συνάδελφο κυρία Σάλτε Μόζε. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει μεν να κοιτάξουμε το συντομότερο δυνατόν να εφαρμόσουμε νομοθετικώς πως τις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σωστή η πρόταση του συναδέλφου Ντάλτον να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να το κάνουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε παρόλα αυτά την ημερομηνία τελικής ψηφοφορίας. Και να φροντίσουμε το θέμα αυτό, γιατί ουσιαστικά το θέμα δεν είναι να τιμωρήσουμε τον οποιοδήποτε, αλλά να φροντίσουμε να υπάρχει μια καλύτερη λύση για τους καταναλωτές των συντομότερων δυνατόν. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να είναι τόσο εύκολο να ορίσει ο νομοθέτης του τι είναι το νόμιμο και τι είναι παράνομο, όπως προτείνει η κυρία Σαλδεμόζε. Φυσικά αυτό θα ήταν ευκταίο στην, στην φάση σύνταξης της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία προφανώς αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία στους, καταναλωτε... στους ε, παραγωγούς από ό,τι θα ήθελε συνήθως ο νομοθέτης. Και έτσι λοιπόν πλήρω αξιοποιήθηκε αυτή η ευελιξία και η ελευθερία. Μην σα πω ότι και έγινε κατάχρηση αυτή σε κάποιε περιπτώσει. Και όταν λοιπόν ξεπερνάμε τα όρια, αυτό είναι παράνομο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει περαιτέρω ορισμό. Απλά θα πρέπει να δράσουν και να αναλάβουν δράση οι αρμόδιε αρχέ. Και ελπίζω λοιπόν οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών να το πράξουν αυτό. Όπω τουλάχιστον έχουν υποδείξει ότι πρόκειται να κάνουν στην παρουσία φάση. Δεν ξέρω να κάνω κάποιε ερωτήσει, ε, κύριε Πρόεδρε, ή απλά να περιοριστώ στα σχόλια. Εγώ θα πρέπει να ομολογήσω με πάσα ειλικρίνεια ότι γνωρίζω εις βάθος μόνο λίγους νομικούς τομείς στους οποίους οι κρατικέ ε, εγκρίσεις για κάποια προϊόντα έχουν α, περιορισμό χρονικό. Αυτό ισχύει για πυρηνικά εργοστάσια και αυτό μου φαίνεται λογικό. Αλλά τώρα γιατί το σύστημα έγκρισης τύπου για οχήματα θα πρέπει να έχει χρονικό περιορισμό 5 έτη δεν το κατανοώ. Αυτό θεωρώ ότι ενδεχομένω να είναι μια γραφειοκρατική υπεραντίδραση, υπερβολική αντίδραση στο σκάνδαλο αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ θα πρότεινα το εξή. Μάλλον το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια ισχύω ε, της έγκρισης ε, θα πρέπει να χρειάζονται πιο πολλοί έλεγχοι και να υπάρχουν διαδοχικές ε, επιθεωρήσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό. Και το γεγονός ότι χρειάζεται ε, ουδέτερα τέλη και αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Να συζητήσουμε βέβαια το πώς θα επιβληθούν τα τέλη αυτά, γιατί δικαίω ε, ε, τέθηκε ένα ερωτηματικό για το κατά πόσον η πρόταση γίνεται προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θεωρώ ότι γενικώ πώ. Ε, η Επιτροπή μας έχει θέσει ένα σωστό πλαίσιο, ένα σωστό χρονοδιάγραμμα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τα πιο ακαθόδη ζητήματα και προσβλέπω στην διεξαγωγή λοιπόν των... Ε, Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν θα έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε το διάλογο με τους ενδιαφερομένους, ε, αλλά αν επιθυμούν να στείλουν τα σχόλιά τους ή τις απαντήσεις τους, ε, μπορούν να το κάνουν γραπτός στέλνοντας στη γραμματεία η οποία θα τα προωθήσει περαιτέρω. Από τους Πρασίνους ο, ο κύριος Τσούλο μήπως έχει ερώτηση. Μια σύντομη παρέμβαση σε σχέση με τα υποθέντα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεμελιώδου σημασία να μιλάμε για ευελιξία, να μην έχουμε ένα σύστημα που είναι εξαιρετικά άκαμπτο αλλά κυρίως για να τηρήσουμε το ίδιο το σύστημα αποτελεσματικό χρονικά, ούτως ώστε α, να ισχύουν είναι οι κανόνες που θα θεσπίσουμε και χρονικά. Είναι ένας τομέας τεχνολογικός που με την πάροδο του χρόνου αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή η πτυχή λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το να δημιουργήσουμε εξαιρετικά κάμπτο σύστημα μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι κάτι αντιπαραγωγικό για όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω το λόγο. Δεν ξέρω ποιος την εκπροσωπεί. Ορίστε κυρία μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη συνεδρίαση και την άκρως ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια που ακούστηκαν και η γενική έγκριση της μεταρρυθμίσεως του συστήματος εγκρίσεως τύπου. Αυτό συνήγαγα από αυτά που είπατε. Εκφράστηκε και αμφιβολίες και ανησυχίες. Οπότε αυτό πάνω το συζητήσουμε. Δύο-τρία σημεία θέλω να θίξω και να προβώ σε δύο-τρει παρατηρήσει που ακούστηκαν. Καταρχά, γιατί γίνεται η μεταρρύθμιση. Προσπαθούμε, ξέρετε, να ξεπεράσουμε τι αδυναμίε του συστήματο. Λειτουργήσε αρκετά καλά το σύστημα. Απέδειξε τα θετικά του στοιχεία, αλλά απέδειξε και τα όρια του. Αναφέρθηκε αυτό σήμερα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί ξανά το σύστημα. Εξετάζουμε το σύστημα στο σύνολό του. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δεν εξετάζουμε διαδικαστικού κανόνε. Με την πρόταση για την έγκριση τύπου εξετάζουμε τα στοιχεία, νομοθεσία περί εκπομπών κλπ. Που αυτό θα καλύψει και αυτά που υπόθηκαν. Εξετάζουμε όλα τα στάδια και όλου του εμπλεκόμενου φορεί δεν θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε λεπτομέρειες του συστήματος χωρίς γενική θεώρηση των πραγμάτων. Πώς γίνεται η σύλληψη, ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου, η παραγωγή του κλπ. Αυτό εν είδη απαντήσεω σε κάποιο σχόλιο που ακούστηκε από πυρογνώμονα, δηλαδή να εξετάζουμε τον όλο κύκλο ζωή του οχήματο. Για αυτόν τον σκοπό εξετάσαμε κάθε παράγοντα και το πλαίσιο εντό του οποίου κινείται κάθε παράγον, ούτω ώστε να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό ε, μελλοντικά προβλήματα και αποτυχίες. Δεύτερον, όμως αφήσαμε ακέρες τις αρχές. Το σύστημα παραμένει αποκεντρωμένο, δεν προτείνουμε κεντρικό φορέα, προτείνουμε έλεγχο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί, όπως είπε και κάποιος εμπειρογνώμων, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα που είναι κεντρικό στα χέρια 28 κεντρικών αρχών να γίνεται εφαρμογή του νόμου ενιαία. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Πρέπει να ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο ο νόμος από όλου. Αυτό είναι ο στόχο τη επισκοπή και του ελέγχου πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τέλο, ο χρόνο που αναφέρθηκε, το χρονικό στοιχείο. Βέβαια, αναγνωρίζουμε πλήρω ότι η πρόταση είναι περιπλοκότατη ω τεχνική και θα πρέπει να διαθέσουμε τον χρόνο εν εξέβρεση καταλήλων λύσεων. Να τονίσω όμω ότι έχουμε μάθει από τη Volkswagen. Έχουμε εξεργαστεί το σύστημα εγκρίσεων τύπου κατά το παρελθόν, μάθαμε και από τη Volkswagen. Δεν πρέπει να δημιουργείται εντύπωση ότι επειδή ξοδεύουμε χρόνο και μήνες συζητώντας τις λύσεις, ότι στο τέλος δεν θα έχουμε κάποια μέτρα διορθωτικά για το σύστημα. Είναι σημαντικότατο να το καταλάβουμε αυτό. Δεν προσπαθούμε να βελτιώσουμε λίγο που, κάτι που δεν λειτουργεί καλά λιγάκι. Θέλουμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν σήμερα. Άρα τίθεται χρονικό θέμα για το κείμενο, είναι πολύ σημαντικό ο παράγον χρόνο. Και από τα σχόλια που άκουσα, τα πιο σημαντικά, πρώτα απ' όλα, το θέμα ε, χρειάζεται οι πληροφορίες οι κατάλληλες για τις διορθώσεις, για τις επισκευές και τη συντήρηση. Θέλαμε να δούμε πώς λειτουργούν οι κανόνες σημερινής. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα ε, και επισκευών, Θέλουμε όμως να λάβουμε υπόψη για διάφορα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και προβλήματα που διωθώνται εύκολα που ίσως να προέρχονται και από κάποιες ασάφειες του κειμένου, οπότε θα δώσουμε κάποια συνέχεια στον αυτό το θέμα της συντήρησης και των επισκευών. Μετά, η οικονομική ανεξαρτησία εθίγει. Εξετάσαμε διάφορες τέτοιες στοιχείες ανεξαρτησίες των κατασκευαστών, των αρχών εγγύσεως τύπου, ε, των αρχών για τις δοκιμές κλπ. Χρειάζεται λοιπόν γενική εποπτεία της αγοράς, αυτό είναι δύσκολο. Θα εξετάσουμε τα στοιχεία μαζί με τους συνομοθέτες. Ποια πρέπει να είναι η αρχή όμως, ότι από πλευρά ποιοτική και οικονομικής και χρηματοδοτήσεως θα υπάρχει ένα τείχο, συνικών τείχο και να μην επηρεάζει μια πτυχή την άλλη. Να μην υπάρχει οικονομική εξάρτηση των τεχνικών υπηρεσιών, των κταίων, παραδείγματο χάρη, από του κατασκευαστέ. Μετά το θέμα των συσκευών που ξεγελούν το σύστημα ελέγχου είναι κάτι άλλο που θα το εξετάσουμε σε άλλη φάση. Είναι στα πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης. Άλλα δύο πακέτα θα ετοιμάσουμε και σε άλλο πακέτο θα εξετάσουμε το θέμα αυτών των συσκευών που ξεγελούν το σύστημα ή defeat devices όπως αποκαλούνται. Αυτά ήταν πιο σημαντικά θέματα που εθήκησαν. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστούμε κύριε Σβιστόσκα. Ο Ντάνιελ Ντάλτον, ο εισηγητής μας τώρα, θα κάνει κάποιες παρατηρήσεις μετά το πέρας αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και τους καλεσμένους μας. Πολύ χρήσιμη συζήτηση. Καταρχήν για το χρονοδιάγραμμα. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν παραθυράκια, κενά και θα παραμείνουν αν δεν υιοθετηθεί η νομοθεσία για να τα σταματήσει. Όσο μακρηγορούμε λοιπόν, όσο χρόνο τριβούμε ε, και παραμένουν τα παραθυράκια, ε, δίνουμε ε, λαβή στου αυτοκινητοβιομηχάνους που και στο παρελθόν ξεγελούσαν να συνεχίσουν να, απατούν, να εξαπατούν. Γι' αυτό θα πρέπει να ολιγορούμε και να διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό τα κακό σκήμενα. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δράσουμε ταχαίως. Ήμουν αρκετά ελαστικός και τροποποίησα τα εσωτερικά μας χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες, αλλά μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και φάνηκε και από τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών. Θα πρέπει να δράσουμε ταχαίως και να διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατό αυτό το θέμα. Κάποια σύντομα σχόλια για τη σημερινή συζήτηση. Ε, η αυτοκινητομηχανία ζήτησε να περικοπεί περιττή γραφειοκρατία. Συμφωνώ. Ούτε και εμεί θέλουμε περιττέ γραφειοκρατικέ διατυπώσει. Αλλά αν δεν προσπαθούσαμε να μα ξεγελάσουν τα κράτη-μέλη, δεν θα βρισκόμαστε στη σημερινή κατάσταση. Προσπάθησαν να μα κοροϊδέψουν μερικά κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά βασικά θέματα, την πενταετία, το χρονικό περιθώριο, με προβληματίζει κάπω. Δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν το πρόβλημα και αυτό προκάλεσε το σκάνδαλο, το χρονικό περιθώριο. Και ίσως ε, ε, για αυτοκίνητα που είναι προσαρμοσμένα σε αναπήρους. Ε, ίσως σε τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίσω πρόβλημα με το πενταετές χρονοδιάγραμμα. Πώς είναι δυνατόν να μην δημιουργηθούν προβλήματα για τα αυτοκίνητα ειδικού σκοπού, αυτά που είναι προσαρμοσμένα για αναπήρικα αμαξάκια, για παράδειγμα. Επίσης, για τα τέλη, με προβληματίζει και η διάρθρωση των ε, τέλων και σφορών Θέλουμε να διαρρήξουμε τον ε, σύνδεσμο μεταξύ των ε, κατασκευαστών αυτοκινήτων και των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου, των ΚΤΕΟ. Θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα υιοθετήσουμε μια λύση ώστε να διαταραχθεί, να διαρριχθεί αυτός ο δεσμός και αν δεν συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνουμε μια εναλλακτική λύση. Τώρα, γιατί τα ανεξάρτητα συστήματα επισκευής ε, και τους ανεξάρτητους ε, επισκευαστές. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε, πώς θα συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τα, για τα γκαράζ επισκευής, ώστε και να μπορούν να το κάνουν εξάρτητα, αλλά να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα τα πνευματικά των κατασκευαστών. Αυτό είναι βασικό θέμα ε, που δεν αφορά μόνο το παρόν και το παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Γιατί τα software αναπτύσσονται ταχύτατα. Ε, στην ψηφιακή εποχή ο ρυθμός πρότεινε ραγδαίος και θα πρέπει να δούμε μια λύση που θα μας εξασφαλίσει και στο μέλλον, σε επόμενα 10-15 χρόνια. Ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει. Και τέλος, για τις ενώσεις, για τα σχόλια της Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών και για αυτά τα συστήματα που ξεγελούν, το είναι παράνομο αν δεν ε, τηρηθούν οι προδιαγραφές ε, ε, καυσέριων. ή αν δεν... Βέβαια, αν απαγορεύσουμε αυτές τις συσκευέ defeat devices, είναι σαν να λέμε ότι όλο το σύστημα είναι προβληματικό. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, αναφέροντας ρητά και κατηγορηματικά τα defeat devices, αυτές τις συσκευέ που ξεγελάνε το σύστημα. Ε, και δίνουν ε, εσφαλμένα στοιχεία για τα καυσαέρια. Θέλουμε να εμποδίσουμε να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Δύσκολη αυτή η νομοθετική πρόταση. Νομίζω ότι είναι σωστή η γραμμή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χρονοδιάγραμμά μας. Θα πρέπει όμως εσωτερικά να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στις συνεδριάσεις μα για το θέμα αυτό, γιατί έχουμε ακόμη πολλές εκκρεμότητες και θέλουμε περισσότερο χρόνο για πιο εκτενή συζήτηση για επιμέρου σημεία στο μέλλον. Ευχαριστώ, Ντανιέλ. Πολύ καλή ανακεφαλαίωση μας έκανες ε, των ε, πιο σημαντικών θεμάτων. Και σίγουρα το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό. Στα αρχές Ιουλίου θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης, ο χρόνος περνάει όμω. Και στα τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Σε λίγα λεπτά θα περάσουμε στην ώρα του νομοθετικού ελέγχου. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Ανεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Μάτες, Προηγουμένως όμως έχουμε μια σύντομη ψηφοφορία. Θα είδατε ότι η γνωμοδότηση της Vicky Φόρντ για το φυλάδιο ε, έχει αναβληθεί, οπότε θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα τη γνωμοδότηση της Βίκης Φόρντ. Θα ψηφίσουμε όμως... Τι γίνεται ξαφνικά φασαρία. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν αθόρυβα. Donc, euh, θα ψηφίσουμε λοιπόν την έγκριση των ε, συστάσεων των συντονιστών της Επιτροπής μας για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2017 οι συντονιστές μήπως ε, θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια πριν ψηφίσουμε. Ανδρές, Βάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί τη αρχή είναι τεχνική μόνο υπόδειξη που έχω να κάνω. Νομίζω ότι ω Επιτροπή Ιστορική Αγορά, με τι πολλέ οριζόντιε αρμοδιότητε που έχουμε, καλύτερα θα κάνουμε να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη σημεία και εκ των προτέρων μεταξύ των πολιτικών ομάδων να συμφωνήσουμε μερικά πράγματα στα πλαίσια της Επιτροπής, γιατί δεν έχει νόημα κάθε πολιτική ομάδα να προσπαθήσει να περάσει τα συμφέροντά της ε, καταρχάς ε, μέσω της Επιτροπής και κατά δεύτερον ε, μέσω της Ολομέλειας. Αυτό στο παρελθόν νομίζω ότι είχε αποδυναμώσει την άποψη της Επιτροπής Εστρικής Αγοράς, αλλά αυτή τη φορά καταφέραμε με την στοχοθετημένη αυτή σύνταξη να τα, βελτι... να τα βελτιώσουμε τα πράγματα. Μάλιστα, δεν θα στερήσω το λόγο, λέει ο πρόεδρος, από κανέναν, αλλά αν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε πάρα αυτά στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε με, τις, ε, με κάρτες. Προτιμάει η γραμματεία. Με την κάρτα ψηφοφορίας λοιπόν θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρω. Έχετε όλοι οι συνάδελφοι τις κάρτες σας μαζί. Έχουμε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί. Πολύ φοβάμαι ότι λείπουν κάποιοι ψήφοι από τη δική μου ομάδα. Έχουμε κάποιους απόντες. Μάλιστα. Έχει καλώς. Πέρασε τη ψηφορίας, αν ψήφισατε όλοι. Πολύ ωραία. toujours ε, Ο Μάρκ πάντα ενθουσιώδης και δυναμικός. Bien, Euh, euh, le vote donc... Euh, Μάλιστα, ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στο νομοθετικό έλεγχο. Ο κύριος Ματές από το ελεγκτικό συνέδριο θα πάρει το λόγο. Chevaillat. Bien, donc je suis heureux d'accueillir euh, Monsieur. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του κυρίου Μάτε, που είναι μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου και υπεύθυνο ε, εισηγητή τη ειδική έκθεση ε, για την εφαρμογή τη οδηγία για τι Υπηρεσίε. Θα ήθελα να σα πενθυμίσω, κύριε Μάτε, ότι οι συντονιστέ τη Επιτροπή ΣΥΜΚΟ αλλά και το σύνολο των ε, μελών της Επιτροπής αποδίδουν ε, ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την ε, παρακολούθηση που γίνεται στην Επιτροπή μας στα θέματα του νομοθετικού ελέγχου και γνωρίζετε ότι όχι μόνο παρακολουθούμε την θέση εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αλλά μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερος το θέμα αυτό. Κύριε Μάτης, λοιπόν, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τα γενικά αποτελέσματα και τις συστάσεις της έκθεσής σας που έχει δημοσιευθεί στις 14 Μαρτίου, σχετικά πρόσφατα, 14 Μαρτίου 2016. Κύριε Μάτας, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να ομολογήσω ότι το ελληνικό συνέδριο έχει δείξει μεγάλη ε, μάλλον χαίρεται ιδιαίτερα που έχετε επιδείξει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τελευταία αυτή έκθεση σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή τη οδηγία για τι υπηρεσίε. Να δώσω κάποια ιστορικά δεδομένα, εν συντομία, κάποιο ιστορικό υπόβαθρο. Πριν από 10 χρόνια και παραπάνω θεωρούταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καλά τα πήγαινε και λειτουργούσε καλά η ενιαία αγορά αλλά η αγορά στις υπηρεσίες αντιμετώπισε πολλά εμπόδια. Και γενικά το επίπεδο εμπορίου σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες μεταξύ των κρατών ήταν ανεπαρκές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρούθηκε ότι είχαμε χάσει και χάναμε πάρα πολύ ε, ΑΕΠ σε ό,τι αφορά τα εμπόδια αυτά. Η αρχική λοιπόν πρόθεση ήταν να υπάρξει η αρχή της προέλευση η ονομαζόμενη, το οποίο τι σημαίνει ότι όταν ένας παραγωγός ε, υπηρεσίας ε, έχει καταχωριστεί και έχει αντιβοτηθεί στη χώρα του και υπόκειται στις ε, σχετικές νομικές διτάξεις, μπορεί λοιπόν να παρέχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά ύστερα για κάποιους λόγους δεν επιλέχθηκε αυτή η λύση. Το 2006 λοιπόν προέκυψε η οδηγία για τις υπηρεσίες και τελικά και από το κρατημέλη να εφαρμόσουν την οδηγία στην εγχώρια νομοθεσία. Ήταν τεράστιο λοιπόν το project το τεράστιο έργο. Από όλες τις οδηγίες ε, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συγκεκριμένη θεωρώ ότι ενδεχομένως να χρειάστηκε το μεγαλύτερο αριθμό τροπολογιών, τροποποιήσεων ε, για την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Τεράστιο όγκο νομοθετήματος ε, θεμητό και λογικό και δεν μας προκαλεί έκπληξη, γιατί καλύπτει τόσα πολλά σημεία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Σκοπός ήταν να αυξηθεί η διαφάνεια, να είναι πιο εύκολη η εμπορία υπηρεσιών. Ήταν μεγάλο το έργο αυτό και είχε πάρα πολύ μεγάλη συνέπειες σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση και την αναθεώρηση της νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Και άρα ορίστηκε περίοδο εφαρμογή τριών ετών, γιατί ήταν και τόσο περίπλοκο και τόσο εκτενέ το έργο αυτό. Είχαν τρία χρόνια λοιπόν στη διάθεσή του τα κρατημέλη για να εφαρμόσουν τι αλλαγέ αυτό. Δέκα χρόνια μετά την ε, οδηγία και 7 χρόνια μετά την λήξη της περίοδου εφαρμογής το ελεγκτικό συνέδριο καλείται να ελέγξει κατά πόσον όντως έχει εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό έχει εφαρμοστεί η οδηγία στα κράτη-μέλη. Και προσπαθούμε συγκεκριμένα να απαντήσουμε στα εξή ερωτήματα. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει σωστά την εφαρμογή τη οδηγία για τι υπηρεσίε, αυτή ήταν η πρώτη υποερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκόλυνε και εφάρμοσε την ε, υλοποίηση της οδηγίας αυτής. Σε τελική ανάλυση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο εν μέρη ήταν αποτελεσματική και αποδοτική ως προς τα ερωτήματα αυτά. Καταρχάς, παρά τη μεγάλη μεταβατική περίοδο τριών ετών, όπως είπαμε, τα πιο πολλά κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να τηρήσουν την προθεσμία. 20 συγκεκριμένα εξ αυτών. Και αυτό οφείλεται σε πολλές αιτίε. Μία από τις αιτίε ήταν ότι το τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο προετοιμασεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία αυτή, κατέστη διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών 11 μήνες μετά την έγκριση της οδηγίας. Η αγγλική εκδοχή ήταν διαθέσιμη 5 μήνες, 4 μήνες πιο νωρίς, αλλά σε όλες τις γλώσσες το εγχειρίδιο, το τεχνικό ήταν διαθέσιμο 11 μήνες αργότερα. Αυτό έπαιξε προφανώς κάποιο ρόλο για την καθυστέρηση της διαδικασίας. Το δεύτερο πράγμα το οποίο ανακαλύψαμε ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, αντιμετώπισε το θέμα της συλλογής δεδομένων αρκετά νωρίς. Δεδομένων τα οποία θα βοηθούσαν για την αξιολόγηση της υλοποίησης της οδηγίας. Ε, τα δεδομένα για την, ε, για την παροχή υπηρεσιών τα πρακτικά για το... τα εμπορικά στοιχεία, τα εμπορικά δεδομένα, ισολογισμοί κτλ. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα χρειαζόντουσαν λίγο παραπάνω ενοποιημένα στοιχεία, λοιπόν, ενοποιημένα δεδομένα για το εμπόριο. Δυστυχώς λοιπόν αυτό δεν έγινε. Το 2014 λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για την ε, συλλογή τέτοιων δεδομένων. Προσπάθησαν να ε, συστήσουν μια εικόνα για το παρελθόν. Αλλά κατάφεραν να φτάσουν μόνο μέχρι το 2012. Δεν υπήρχαν λοιπόν ε, αδιάσυστα στοιχεία για να υπολογιστεί πόσο έχει αυξηθεί το εμπόριο στις υπηρεσίες μετά την εφαρμογή της οδηγίας. Έλειπαν στοιχεία δηλαδή ε, μέχρι το 2012. Τώρα, το κατά πόσον έχουν παραμείνει τα εμπόδια στην εμπορία υπηρεσίων. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και πολλές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι εξακολουθούν να, υφαρ, να υφίστανται τέτοια εμπόδια. Αυτό προκύπτει από μία έρευνα το 2011 και από τις ε, επαφές που είχαν οι ελεκτές μας με τα κρατημέλη κατέληξαν στη Γενική Συμφωνία ότι δεν υπήρξε επαρκές follow-up από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινή αυτής ε, διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλη του 2015 δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον έγγραφο για τα αναπομείναντα ε, εμπόδια. Και το ποιες είναι οι δυνατότητες εξάλληψης των εμποδίων αυτών και τι συνέπεια θα είχε αυτό στην αύξηση του ΑΕΠ στην Ένωση. Η εικόνα η οποία αποκρισταλώθηκε από αυτό το πολύ ενδιαφέρον έγγραφο είναι η εξή. Ε, χοντρικά. Ότι μετά την υλοποίηση, ακριβώς μετά την υλοποίηση, υπήρξε κάποια πρόοδος, αλλά αυτή η πρόοδος στη συνέχεια ανακαμφθήκε μεταξύ 2012 και 2014 δεν σημειώθηκε ουσιαστικά πρόοδο. Κάποιες χώρες εξάλληψαν περαιτέρω εμπόδια, έκαναν παραπάνω βήματα και αυτές ήταν κυρίως χώρες όπου υπήρχε υποστήριξη ισολογισμού ε, πληρωμών ε, λόγω μνημονίων ή υπήρχε πρόβλημα λόγω ε, εθνικής, εθνικού χρέους στις υπόλοιπες χώρες ουσιαστικά η τάση ήταν αντίστροφη και τελικά ο καθαρός αντίκτυπος των εξελίξεων μεταξύ 2012 και 2014 στο ΑΕΠ, στο επίπεδο ΑΕΠ υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μόνο 0,1% ποσοστό αντίστοιχο του ΑΕΠ. Όταν υπολογίστηκε όμως ε, πόσο μεγαλύτερο ήταν το πεδίο εφαρμογή, ε, καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι ενδεχόμενη αύξηση στο επίπεδο ΑΕΠ με εξάλληψη περαιτέρω εμποδίων θα μπορούσε να φτάσει στο 0,8 έως 1,8%. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 0,1% το οποίο είχε πραγματοποιηθεί. Το γεγονό λοιπόν είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια σε τι οφείλεται τώρα αυτό και ποια είναι η δική μας η εκτίμηση. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρκετά απρόθυμη να εκκινήσει ε, νομικές διαδικασίες. Αυτό σε κάποιο βαθμό οφείλεται στη διάρκεια, τη μεγάλη διάρκεια των ε, νομικών αυτών διαδικασίων και υπήρχε και γενικώ έλλειψη εμπιστοσύνη στην ε, σχετική νομοθεσία. Αυτό μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει εκτάσει πιο επακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της αναλογικότητας, το οποίο χρησιμοποιείται από κάποια κράτη-μέλη ως επιχείρημα για τη διατήρηση κάποιων εμποδίων. Και εδώ πέρα τα πράγματα περιπλέκονται λίγο, γιατί αφενό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι μόνο το ΔΕΚ μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα για την αναλογικότητα. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν και να ε, καταγγείλει τις περιπτώσεις αυτές στο 10. Άρα, ύστερα, χρησιμοποιήθηκαν ε, τη δικασία που παραβάζει αρκετά σπάνια. Ουσιαστικά, μία μόνο περίπτωση κατέληξε στο δικαστήριο. Αντί να εφαρμόσει λοιπόν και να κινήσει τέτοιε διαδικασίε επί παραβάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε στον νέο μηχανισμό σε μεγάλο βαθμό. Το EU Pilot, όπω ονομάζεται. Πρόκειται για ένα σύστημα διεξαγωγή άμεσου διαλόγου με τα κρατημέλη, χωρί όμω να ανακοινώνεται το αντικείμενο του διαλόγου ή το αποτέλεσμα του διαλόγου. Είναι αυστηρά εσωτερική διαδικασία αυτή του διαλόγου για να επιληθούν κάποια ζητήματα. Άρα, συνολικά το EU Pilot ή οι διαδικασίες επί παραβάση, όλα αυτά παίρνουν χρόνο, παίρνουν πολύ χρόνο και δυστυχώς η οι διαδικασιες επι ολα αυτα παιρνουν χρονο Επιτροπή δεν ακολουθεί, δεν παρακολουθεί συστηματικά τέτοιες υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Ξέρουμε ότι σε ένα χρονικό σημείο μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2014, αν δεν κάνω λάθος, η μέση διάρκεια εκκρεμουσών υποθέσεων ήταν 20 μηνών. Εκκρεμούσε, σε τονίζω, υποθέσεις τέτοιες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Από άλλες δε ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις διαδικασίες επί παραβάση που υπάγονται στις πολιτικές εσωτερικής αγοράς και όπως δήλωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτός όμως ο χρόνος, αυτή τη μέση διάρκεια, έρχεται σε 30 μήνες. Αν είναι λοιπόν κανείς μια μεγάλη εταιρεία, ένας μεγάλος όμιλος, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να περιμένει ένα χρόνο. Αν είναι κανείς μικρομεσαία επιχείρηση, αυτού, δεν ε, μπορεί να το ε, εντάξει κανείς στις εργασίες τους. Αν παίρνει τρία χρόνια η διαδικασία αυτή, προφανώς αποθαρρύνεται και η μικρομεσαία επιχείρηση. Και αυτό έχει φυσικά και επιπτώσεις και στον καταναλωτή, ο οποίος ενδεχομένω να ήθελε να δείξει ένα τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα. Στη συνέχεια, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να δείξει και λίγο πιο ανοιχτό πνεύμα σε ό,τι αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τις, ε, την οδηγία για τις υπηρεσίες και στο EU Pilot και σε μία διαδικασία που παραβάσει. Υπάρχουν, κάποια υπάρχουν ανακοινώσεις τύπου στην αρχή και στο τέλος, αλλά το τελικό έγγραφο ουσιαστικά δεν δημοσιεύεται και δεν δημοσιεύεται ουσιαστικά και στο τέλος της διαδικασίας το πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα το οποίο οδήγησε στη διαδικασία να παραβάσει. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ε, τομέα αυτό βοηθούσε για να δημιουργηθεί μια κοινή διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί θα, θα θέλαμε να ξέρουμε τι έγινε σε μια άλλη χώρα, για παράδειγμα. Γιατί η απάλληψη τέτοιων εμποδίων Ουσιαστικά, α είμαστε ειλικρινεί, έχει να κάνει με προστατευτικά μέτρα. Ο εμπόδια και προστατευτισμός ουσιαστικά το ίδιο είναι. Άρα, όσοι προτίθενται να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν την οδηγία για τις υπηρεσίες ε, απελευθέρωση του εμπορίου, δηλαδή, θεωρώ ότι θα βοηθούνταν αν ήξεραν τι ακριβώς συνέβη σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάξαμε το θέμα αυτό. Ποιες είναι λοιπόν οι συστάσεις μας. Νομίζω ότι αναφέρεται με ορισμένε εξ αυτών, αλλά να πω και δύο λόγια παραπάνω. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει αυτή την αμοιβαία διαδικασία αξιολόγηση, θα πρέπει να παρακολουθεί με πιο μεγάλο σύστημα το τι θα γίνει σε όλη τη χρονική διάρκεια από ό,τι έχει συμβεί έως τώρα. Και πιστεύουμε επίσης ότι η διάρκεια της διαδικασίας και στα πλαίσια του EU Pilot και στα πλαίσια της διαδικασίας επιπαραβάση ε, θα έπρεπε να μειωθεί γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πραγματικά απαθαρρύνει πάρα πολύ κόσμο από το να καταγγείλει τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνονται και καταγγελίες στο ΔΕΚ. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή μόνο μία υπόθεση να έχει φτάσει στο δικαστήριο είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί και μας απασχολεί. Άλλες συστάσεις θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να γίνονται σεβαστοί οι χάρτες για τα σημεία ενιαίας επαφής. Εδώ πέρα, οι διάφορες χώρες ακολούθησαν διάφορες διαφορετικές διαδικασίες. Σε κάποιες χώρες πήγε καλά αυτό, σε κάποιες άλλες δεν πήγε τόσο καλά. Και θα πρέπει φυσικά να βελτιωθεί η κατάσταση. και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσουν προκειμένου να υπάρξει πρόοδο στο θέμα αυτό. Υπάρχει το θέμα της περίοδου αναστολής, standstill, όταν ε, η χώρα θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, την οδηγία για τις υπηρεσίες. Στην παρούσα φάση τα κρατημέλη έχουν ε, υποχρέωση να αναφέρουν α, τις αλλαγές αυτές, αλλά δεν υποχρεούνται να ζητήσουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των άλλων κρατών μελών. Άρα προτείνουμε τέτοια περίοδος standstill να εφαρμοστεί και στην ε, περίπτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, όπως ισχύει και σε άλλους κλάδους. Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, υπάρχει το SWEEP ένα σύστημα όπου ελέγχονται οι ιστοσελίδε των διαφόρων παρόχων για να μην υπάρχουν διακριτικέ ε, συμπεριφορέ κτλ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η υπηρεσία για τις οδηγίες να συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα SWEEP αυτό. Γενικώ πώς θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά την ε, καθοδήγηση για την ε, υλοποίηση τέτοιων πολυσύνθετων ε, καινούριων οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο γρήγορη, να είναι πιο ταχεία στις αντιδράσεις της, για να παρέχει εγχειρίδια, ενημερώσεις κτλ. Και θίξαμε ήδη και το θέμα των κατάλληλων και σωστών στοιχείων. Αυτό θα πρέπει να εισαγάγεται νωρί, ε, εγκαίρω στην νομοθετική διαδικασία, όχι τόσο αργά όσο έγινε στην συγκεκριμένη οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε όλε μα τι συστάσει, εκτό από αυτή που έχει να κάνει με το EU Pilot. Υπάρχει απόφαση δε του ΔΕΚ που ε, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπιστευτικό και απόρριτο χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει στα πλαίσια του EU Pilot. Αλλά το δικαστήριο είπε ότι αυτό ισχύει για την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όχι μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Προφανώ, ναι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπάρχει απόρριτο χαρακτήρα. Αλλά στο τέλο, όταν πλέον έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν μπορεί να δημοσιεύεται το αποτέλεσμα αυτό. Άρα, Συνολικό πώς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο ενεργή σε ό,τι αφορά θέματα εφαρμογής της οδηγίας. Αλλά, όπως σημείωσε το ελεκτικό συνέδριο, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε πιο ενεργή στάση και έτσι ξεκίνησαν και παρακολουθήθηκαν πιο πολλές διαδικασίες μη συμμόρφωση από ότι στο παρελθόν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα ενθαρρύνει το γεγονό ότι η νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά που εγκρίθηκε το Οκτώβριο του 2015 έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με πολλά ζητήματα τα οποία έχουν ε, εφαρμογή και στην οδηγία για τι υπηρεσίε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σα και εγώ και οι συναδελφοί μου για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ. Όσοι θέλουν το λόγο παρακαλώ να το δηλώσουν. Ο Αντρέας Σφάμπ είναι ο πρώτος στον κατάλογο των αγορητών παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αξιότιμο εκπρόσωπο του ηλεκτρικού Συνεδρίου για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Καταρχάς, θα ήθελα από πλευρά αρμοδιότητας να θέσω και το εξή ερώτημα. Το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, τι δουλειά έχει να μπλέκεται στο πολιτικό σκέλος της αξιολόγησης της υπηρεσίας ε, για τις ε, υπηρεσίες. Αλλά κοιτάξτε, πάντα είναι καλό να συζητάμε την οδηγία για τις υπηρεσίες, οπότε θεωρώ ότι καλό είναι το γεγονός ότι το συζητάμε αυτό και ότι συζητάμε το τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και Ευρωπαίος νομοθέτης, εμείς δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνουμε για να φροντίσουμε να είναι καλύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε επίπεδο κρατών μελών. Και θεωρώ ότι έχουμε πραγματικά τον ίδιο στόχο, κύριε Μάτε. Πιστεύω ότι ήταν επικίνδυνο αν θέταμε την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες ως ε, σημείο αναφοράς για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε εθνική νομοθεσία, γιατί λίγες είναι οι οδηγίες οι οποίες έχουν ελεγχθεί τόσο πολύ ως προς την υλοποίησή τους. Εσείς δυστυχώς καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα και πιο γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι γενικά είναι πολύ μεγαλύτερε ε, οι ελλείψει ό,τι αφορά την εφαρμογή οδηγιών στην εθνική νομοθεσία από ότι αυτά που αναφέρεται ε, για τη συγκεκριμένη οδηγία. Θα θυμάστε πριν από κάποιους μήνες, κύριε Πρόεδρε, είχαμε εδώ τον Μάριο Μόντι, ο οποίος ε, δήλωσε ρητά ότι θεωρεί ότι ένα βασικό μέσο για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια είναι να έχει σωστές αρμοδιότητες ε, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, όπως και ο Επίτροπος Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να έχουμε ε, πιο γρήγορες διαδικασίες αντίδρασης και καταγγελία στο ΔΕΚ, το οποίο δεν επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί Θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα θεσμικό δίλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τοποθετηθεί ε, εξίσου αυστηρά εναντί των κρατών μελών όπως θα επιθυμούσατε εσείς τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Και σε ό,τι αφορά τους Πολωνούς, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ε, η αποφασιστική αντίδραση που θα θέλαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν ένα θεσμικό δίλημα. Θα ήθελα να θέσω τρει ερωτήσει, για τρει συστάσει, μάλλον, για την πρώτη σύσταση καταρχά Να θέσω μια ερώτηση. Δεν είμαι τόσο βέβαιο κατά πόσον ε, στο σημείο αυτό το ελεκτικό συνέδριο παραπλανήθηκε κάπω από τα κρατημέλη, γιατί σε περίπτωση ελλείψεων ε, και καθυστερήσεων σε θέματα υλοποίηση στην εθνική νομοθεσία, πάντα τα κράτη-μέλη προτιμούν να ρίξουν ε, το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Βρυξέλλες. Αλλά δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος κατά πόσον πραγματικά η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του εγχειριδίου ε, οφείλεται σε ζητήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη δικαιολογία αυτή που πλευρά των κρατών μελών. Η τρίτη σύσταση σε ό,τι αφορά τις ε, γραμμή 37 έως 42 σε ό,τι αφορά την ε, εννοείται την ε, προκαταρτική δημοσίευση ή τον των δημοσίευση. Γιατί εδώ θεωρώ ότι ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα. Και μόνο σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, των, του πίνακα ασυσχετισμού, ε, εδώ πέρα είχαμε ζητήματα και το Κοινοβούλιο νομίζω ότι υποστηρίζει στην προκειμένη περίπτωση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπα και αυτό και στην αρχή ότι μου φαίνεται περίεργο το ελεκτικό συνέδριο υποδεικνύει στο νομοθέτη το τι πρέπει να κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το συμφέρον και αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό στόχος. Ευχαριστούμε κύριε Σουβάπη. Κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ελεκτικό Συνέδριο και τον κύριο Μάτες για την ε, καλή αυτή παρουσίαση και για όλα όσα μας ε, είπε. Υποστηρίζω την τοποθέτηση ότι η υπηρεσία, ότι η ιστορική αγορά σε ό,τι αφορά την υπηρεσία θα έπρεπε να λειτουργεί καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα εμπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν. Όλα τα εμπόδια που προκαλούν διακριτική μεταχειρίση. Και συμφωνώ ότι σε κάποιους τομείς ε, της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν λειτουργεί σωστά η ενιαία αγορά και θεωρώ ότι εδώ πέρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό τη ενιαία αγορά και όντω τα κρατη σε κάποιες ε, περιπτώσεις εισαγάγουν δικαιολογημένα ή και αδικαιολόγητα κάποιες, ε, κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά την ε, δραστηριοποίηση στο εμπόριο. Αφετέρου, σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αρκετά μονομερής προσέγγιση και μέθοδος εργασίας. Στην Ουγγαρία υπάρχει για παράδειγμα ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους παρόχους κάποιων υπηρεσιών να παρέχουν υπηρεσίες ενώ η δραστηριότητα αυτή δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Και εδώ ο στόχος ε, είναι να βοηθηθούν για παράδειγμα οι οικογένειες ε, που ζουν στη φτώχεια. Αυτό το πρόγραμμα έχει στεφτεί με επιτυχία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε μια προσέγγιση που δεν δίνει κάποια προνόμια και προφανώς ε, σημαίνει και κάποια τακτική μεταχείριση κατά κάποιων άλλων παρόχων. Ε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο σκοπός ήταν διαφορετικό. Δεν ε, πρόκειται για κερδοσκοπικές δραστηριότητε, τονίζω. Καλό θα ήταν λοιπόν όταν εκείνη η διαδικασία επιπαραβάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ήδη ελέγξει ποιος είναι ο στόχος των δράσεων του εκάστοτε κράτους μέλους, γιατί στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο πολύ ζημιά προκάλεσε. Προφανώς υπάρχουν και επιχειρήσεις και εταιρεία, εταιρείες που ασκούν έντονες δραστηριότητε λόμπι, αλλά σε γενικές δρομές δεν θα πρέπει να περιορίζεται υπερβολικά η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην φοράμε παροπίδες και θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό που έχει η αγορά αυτή. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κάθμι Στάιλερ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και τους προλαλήσαντες. Όταν συμφωνήσαμε σε κάποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε συμφωνήσει σε κάτι πριν από μια δεκαετία. Και μάλιστα οι κανόνες δεν εφαρμόζονται με τον τρόπο που είχαμε συμφωνήσει. Και αυτό είναι πρόβλημα και αντιμετωπίζουμε μεγάλη πρόκληση. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε εδώ με τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις καταθεντήρες γραμμές και τις ολιγορίες, ε, άντλησε κάποια συμπεράσματα, έμαθα το μάθημά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί μέσα 11 μήνες ε, ε, βγήκαν οι κατευθυντήριες γραμμές, οπότε μένω μόνο δύο χρόνια για την εφαρμογή, είναι τριετής η περίοδος. Μιλήσατε 20, ε, για 20 με 30 μήνες ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες στα δικαστήρια. Και ε, η Ουγγαρία έχει άλλου προκλήσεις. Ε, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε με την δικαστική υπόθεση που αφορούσε την Ουγγαρία και ποια ήταν η συνέχεια που δόθηκε. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των δεδομένων, Είχαμε λάβει μια συμφωνία, είχαμε καταλήξει μια συμφωνία το 2006, τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια. Είμαστε μια επιτροπή αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο. Δεν πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς την συνεργασία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κάτι που θα μας διευκολύνει στην ανταλλαγή των πληροφοριών και δεδομένων. Συμφωνείτε. Επίσης μιλήσατε για το EU Pilot που δεν δημοσιεύθηκε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το προωθήσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Τέτοιου είδου ε, συνεργασία χρειαζόμαστε με το ηλεκτρικό συνέδριο. Και όπως είπατε κι εσείς, μόνο το 0,1 του ΑΕΠ ε, ενώ θα μπορούσαμε να αυξήσουμε στο 1,8 την επιρροή ε, για την ανάκτηση. Νομίζω ότι με συνεργασία μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την αλλαγή που χρειαζόμαστε στην ευρωπαϊκή οικονομία ε, εξαιτία τη ε, αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ε, κλάδων. Ευχαριστώ, Κάθριν. Αν δεν υπάρχει άλλο κανεί. Α, συγγνώμη, κυρία Τούν. Mm. Ευχαριστώ. Μια και έγινε μια πολιτική ανάλυση του τι συνέβη στην ε, ενιαία αγορά με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ε, θα ήθελα να μου πείτε αν το ελεκτικό συνέδριο εξέτασε καθόλου τη κατάσταση στο διασυνοριακό εμπόριο. Για παράδειγμα, τι κονδύλια ε, χάνουμε εκεί. Μιλήσατε για την απασχόληση. Δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εκεί θέση εργασίας. Αν είχαμε μια εναρμόνιση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, στην εσωτερική αγορά. Και αν ε, είχαμε πιο εύρυθμη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών και δεν είχαμε τόσο ανυπέρβλητα εμπόδια για τους εμπορικούς τελεστές. Θεωρείτε ότι θα είχαμε πρόοδο σε τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ, Ρόζα. Ο κύριος Στέφαν Εκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Στέφανα, συγγνώμη. Η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ κρίσιμη στον τομέα των υπηρεσιών, όπως επισημάνατε κι εσείς. Είναι σαφές ότι δεν αξιοποιούμε στο έπακρο το δυναμικό μας στον τομέα των υπηρεσιών. Ερωτώ λοιπόν. Ε, μιλήσατε μόνο για την οδηγία της υπηρεσίας, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν έχει γίνει απελευθέρωση όλων των υπηρεσιών στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Ερωτώ λοιπόν, καλύπτεται και εκείνες τις υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική οδηγία για τις υπηρεσίες. Και ναι, πώς τις αντιμετωπίζετε, τις συνυπολογίζετε σε αυτό το δυναμικό ε, για το ΑΕΠ. έγινε μια, ένας υπολογισμός, μια εκτίμηση του δυναμικού για την ανάπτυξη στο ΕΠ ε, από την ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια και να υποβάλω και μία ερώτηση. Σας ευχαριστώ θερμά, όχι μόνο για τη σαφήνεια της ε, εισαγωγής σας και της παρουσίασης σας, αλλά και για την ε, ευκρίνεια της έκθεσής σας που είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστη και εύληπτη, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο σε τόσο περίπλοκα ζητήματα γιατί το ελεκτικό συνέδριο, όπως ξέρουμε, είναι ένα θεσμικό όργανο που είναι πολύ σχολαστικό, δίνει εντελεχείς αναλύσεις. Πάντως ήταν πολύ ευχάριστη και ανάγνωστη η έκθεσή σας. Όπως είπατε και εσείς και επισήμαναν και οι συνάδελφοι, ασχολούμαστε κυρίως με τις δυσκολίες εφαρμογής της οδηγίας αυτής και με του τι συμβαίνει όταν η κατάσταση χωλαίνει στην εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Και συμφωνώ με τον Ανδρέα Σουαβ ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμωνα στο θέμα αυτό. Θέλει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά το έργο της ε, είναι πολύ δύσκολο. Είπατε ότι οι διαδικασίες επί παραβάση δεν ε, πάνε και πολύ καλά, γιατί είναι χρονοβόρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διστάζει να τις ε, αμφισβητήσει. Είπατε ότι προσπαθήσατε στις συστάσεις αναχώρα να τα συμπεριλάβετε αυτά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μάλιστα και η πατρίδα μου η Γαλλία στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των αριθμισμένων κλειστών επαγγελμάτων εμπίπτει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το στόχο. Βέβαια, οι συστάσεις αναχώρα έχουν μια πιο πολιτική διάσταση. Και λέτε, ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια στον ΑΒ τομέα. Ε, έχουν πιο πολιτικό χαρακτήρα αυτές οι συστάσεις χώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βέβαια, το ότι υποβάλλει τις συστάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα γίνουν δεκτέ. Γιατί είδατε στη συστάσει για το 2014 ότι το 2015 δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί. Θεωρώ, εξού ερώτηση, ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει δύο επίπεδα. Το άμεσο επίπεδο, τα κακοσκήμενα, ε, γιατί βλέπουμε που υπάρχουν ανεπάρκειες και τι πάει στραβά. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, πιο απότερο, ε, που αφορά το πώς θα πείσουμε τα κρατημέρια θα πρέπει να γίνει κάπως ε, συγκεκριμένο τρόπο, γιατί κάτι τέτοιο προποθέτει μερικές φορές ε, δύσκολες ε, μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι εύκολο να ρυθμιστεί το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων, των ρυθμισμένων επαγγελμάτων, γιατί προκαλούνται μερικές φορές πολύ συντεχνιακές ε, και έντονες αντιδράσεις. Ίσως με τις στάση αναχώρα σταδιακά και με το χρόνο θα αλλάξει η νοοτροπία. Και όταν έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, χρησιμοποιώντας την αρχή της επανάληψης, ε, η επανάληψη είναι μήτερη της μάθησης, ίσως έτσι έχουμε κάποια ε, αλλαγή και κάπως κινήσουμε τα πράγματα. Έχουμε, έχετε δύο λοιπόν εργαλεία, τις διαδικασίες παραβάση και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο εργαλεία είναι μάλλον συμπληρωματικά ή μήπως αποκλείονται. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκ παραλλήλου ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για την έκθεση και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Όσον αφορά αυτό το εγχειρίδιο, τον οδηγό, η οδηγία περιπηρεσιών ακολούθησε κάποια νέα προσέγγιση. Καλύφθησαν διάφοροι τομείς. Στο τέλος αυτό το εγχειρίδιο ήταν χρήσιμο. Αυτό ανακαλύψαμε. Εξετιμήθη από τα κράτη-μέλη. Άρα έπαιξε το ρόλο του. Παίζει ρόλο όμως και ο χρόνος πέραν το χειρίδιο. Όσον αφορά τα στοιχεία, κάτι που ανέφερε ο κύριος Φαμπ. Όταν έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξασφάλιζε ότι συναλέγησαν τα στοιχεία, είχα υπόψη μου στατιστικά στοιχεία για τις εμπορικές υπηρεσίες που θα καλύπτονται από την οδηγία περί υπηρεσιών. Τα στοιχεία για, τα εμπορικά, ε, για τον εμπορικό τομέα που συλλέγει τα κάτι μέλη ε, εμπεριέχουν στοιχεία για τις υπηρεσίες. Εξαγωγή τουριστικών υπηρεσιών, Φερρυπίν. Είναι κάτι διαφορετικό. Συμπεριλαμβάνονται και άλλα πράγματα. Για να έχουμε σαφή εικόνα να ξέρουμε κατά πόσο η οδηγία Περιπηρεσιών βοήθησε για την αύξηση του εμπορίου υπηρεσίε χρειάζονται βασικά στατιστικά στοιχεία. Δυστυχώς η συλλογή αυτών δεν οργανώθηκε εξ αρχής. Δεν θα απαιτεί το και μεγάλη προσπάθεια πλευράς των μελών. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται. Απλώς έπρεπε να παρουσιαστούν ε, με άλλη ομαδοποίηση. Στο τέλος του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε ότι πρέπει να γίνει αυτό και το επεξεργάζεται το θέμα, αλλά κάπως καθυστερημένα κινήθηκε. Για τα σχόλια του κύριου Σβάμπ, του κυρίου για τη σύστασή μας προς τους νομοθέτες. Δεν είναι έλεγχο συμμόρφωση ο έλεγχο που κάνουμε. Αν κάναμε έλεγχο συμμόρφωση, θα κοιτάζαμε κατά πόσο κάποιοι συγκεκριμένοι κανονισμοί, κάποια νομοθεσία ακολουθείται ή όχι αν όλοι συμμορφώνονται με αυτά που αναφέρονται εκεί. Εδώ ελέγχουμε την επίδοση, αξιολογούμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους. Αν υπάρχουν ελλείψεις και κενά, όσον αφορά αυτό που αναφέρεται και θεσπίζεται σε κάποια νομοθεσία, το παρουσιάζουμε, αυτό κάναμε. Η υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν περί επικειμένων αλλαγών για θέματα οδηγία υπηρεσιών είναι κάτι που υφίσταται. Προβλέπεται την νομοθεσία. Αντίθετα από άλλου τομεί όμω τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ενώσεω που προβλέπουν μία περίοδο αναστολής αν θέλετε στα, στασιμότητας όπου μπορούν να σχολιάσουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει για την οδηγία υπηρεσιών. Εμείς προτείνουμε αυτό που είναι συνηθισμένη πρακτική σε άλλους τομείς της νομοθεσίας και θέλουμε αυτό να ισχύσει και για την οδηγία περιπηρεσιών. Δεν είμαστε ρίζοσπαστικοί. Είναι μια πρακτική που ακολουθείται συνηθισμένη σε άλλους τομείς. Τώρα, αν αξιολογήσαμε το θέμα του ΦΠΑ. Όχι. Για διάφορους λόγους εδώ ασχολούμεθα με την οδηγία περιπηρεσιών. Δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. Έχει σημασία πράγματι ο ΦΠΑ. Τι είδαμε ότι οι επιχειρήσεις συχνά θεωρούν το οργανισμό για το ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ότι είναι περιπλοκότερος από τους κανόνες που αφορούν το εισόδημα και τα κέρδη. Ε, εμείς θα περιμέναμε ότι ο φόρος εισοδήματο είναι κάτι πιο περίπλοκο από τον ΦΠΑ. Αυτό θεωρούν όμω οι εταιρείε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Συμφωνώ ότι η διαφοροποίηση στον ΦΠΑ και στους κανονισμού για το ΦΠΑ δυσχεραίνει τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να παρέχουν εύκολα υπηρεσίε. Το κόστος της συμμορφώσεως ε, είναι κάτι σημαντικό. Δεν το ελέγξαμε αυτό. Αυτό αφορά περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε αυτούς του υπολογισμούς. Εμείς αξιολογούμε εκ των υστέρων αποτελέσματα μιας πρωτοβουλία. Σαν οικονομολόγος και από αυτά που έμαθα από τον έλεγχο επιβεβαιώνω ότι πράγματι η περιπλοκότητα και η διαφοροποίηση στην ομοθεσία του ΦΠΑ στα διάφορα κράτη-μέλη είναι ένα πρόβλημα και επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο, σίγουρα, κυρίως μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. γιατί διαλέξαμε την, ε, την οδηγία υπηρεσιών για να ελέγξουμε. Πρόσφατα διεύρυνε το λεκτικό συνέδριο το θεματολόγιο που καλύπτει. Παραδοσιακά οι ελεγκτές εστιαζόταν επί ελέγχων χρηματοπιστωτικών και συμμορφώσεως χρηματοπιστωτικών ελέγχων αν είναι τα λογιστικά βιβλία εντάξει, συμμόρφωσης αν έχουν εφαρμοστεί σωστά οι κανονισμοί. Το λεκτικό συνέδριο όλο και περισσότερο κινείται προς αξιολόγηση επιδόσεων. Εκεί αξιολογεί κανείς κατά πόσο κάποιο νομοθέτημα και κάποιες πολιτικές πετυχαίνουν τους στόχους τους. Γι' αυτό επιλέξαμε την οδηγία περί Πρόσφατα είχαμε κάνει και έναν έλεγχο του κατά πόσο εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεσματικά στατηγική καταπολέμηση απατών στον τομέα του ΦΠΑ και έχουμε και άλλες πολλές ειδικέ εκθέσεις για διάφορους τομείς. Ζητώ συγγνώμη αν λησμόνησα κάποιες ερωτήσεις. Ας, ας μη σχολιάσω μια κρεμούσα υπόθεση. Δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία της υποθέσεως. Το παραθέσαμε ως παράδειγμα. Είναι το μόνο ζήτημα που παρεπέμφθη στο ΔΕΚ. Θα σταματήσω εδώ, δεν θα σχολιάσω. Ας δώσω το λόγο στο συνάδελφο να απαντήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Στάιλερ, ρωτήσατε ποια είναι η σημασία τη ηλεκτρονική κυβερνήσεω. Επισκεφθήκαμε διάφορε χώρε και είδαμε ποικιλομορφία όσον αφορά τη φιλοδοξία που υπάρχει για τα νέα σημεία επαφή. Και γι' αυτό κάναμε σύσταση ότι κάτι μέλη θα πρέπει να σεβαστούν το, τη χάρτα για τα σημεία επαφή επιθελοντικής βάσεως επί του παρόντος, αλλά θέλουμε να σεβαστούν το πιο φιλόδοξο επίπεδο απαιτήσεων που καθορίζει η Οδηγία Υπηρεσιών δεν είναι πολύ στεναρή όσον αφορά τι απαιτήσει τη και η ηλεκτρονική δυνατότητα διεξαγωγής ε, διοικητικών υποθέσεων είναι κάτι σημαντικό. Α, για την υπόθεση την Ουγγρική. Στο σημείο, στο κεφάλαιο 6 της εκθέσεως, στο τετράγωνο υπαριθμών 6 περιγράφεται, δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο αναφοράς, ο αριθμός αναφοράς, σελίδα 38 του αρχικού εγγράφου σε μορφή Word και μετά είμαστε στο τετράγωνο 6 στο έγγραφο στη μορφή PDF. Παναφερόμαστε στην Ουγγαρία. Καλώς. Πριν εκπνεύσει ο χρόνος μας για το θέμα, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι είναι θέμα, είναι δική της εργασία και ήταν στόχος μέχρι τώρα και ο Γιούργεν. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα ήθελα απλώς να εστιαστώ επί μίας συστάσεως την υπαριθμόν 7 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Όλες οι άλλες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν δεκτές, άρα δεν χρειάζεται η συζήτησή τους εκ νέου. Η σύσταση λοιπόν υπαριθμών 7 περιέχει δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα για τα EU Pilots. Να υπενθυμίσω ότι όταν διεξήχθη ο έλεγχος τέλος του περασμένου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 80 τέτοια EU pilots πιλωτικά προγράμματα όσον αφορά την οδηγία ε, υπηρεσιών. Αυτό σας δείχνει ότι είχαμε 80 τέτοια EU pilots, μια ε, δικαστική υπόθεση που πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα ε, με τα κράτη-μέλη, να τα λύνουμε εκ των προτέρων, ανάντι. Είναι σαφές για μας ότι το EU Pilot ανοίγει ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη τα δέχονται, τα EU Pilots θέλουν να συμμετέχουν. Πιστεύουμε θεσμικά ότι ίσως γίνει πολύ δύσκολη κατάσταση όταν κάθε τέτοιο πρόγραμμα EU Pilot εκτίθεται στο κοινό. Τα κράτη-μέλη ξαφνικά αισθάνονται ότι δεν έρχονται σε επαφή μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να να λυθεί ένα θέμα, θεωρούν ότι θα κατηγορηθούν, θα δεχτούν επίθεση. Γι' αυτό έχουμε κάποιες, κάποια επιφύλαξη και λέμε ότι τα μοδοποιημένα στοιχεία για τα EU Pilots θα έπρεπε ε, να δημοσιεύονται δίνουμε ενημερώσεις περί τίνος πρόκειται και τι βρίσκεται στην οδηγία και τι στο εγχειρίδιο για την εφαρμογή της οδηγίας. Αυτά χρησιμοποιούμε εμείς όταν κινούμεθα οι πληροφορίες που είναι κρίσιμες για κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται εκεί, είναι διαθέσιμες. Αυτό έχω να πω έτσι στα 7, δηλαδή για να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των EU Pilots. Αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα για το ίδιο το εργαλείο EU Pilot. Σας ευχαριστώ ξανά για την συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν θέλω να δώσω αρνητική εικόνα για κάτι που εμφανίστηκε σαν πολύ θετικό. Ε, αυτά έχω να πω μέχρι τώρα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως. Αλλιώς θα θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτησή μας. έχετε κάτι να πείτε μήπως. Κάτι που θυμείτε να πείτε. Όχι, τίποτα από στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέχασα να πατήσω στην ερώτησή σας στις συστάσεις αναχώρα. Εδώ λέγουμε ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε ότι είμαστε πιο, α, πετυχαίνουμε καλύτερα στόχους. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και συστάσεις αναχώρα. Όταν ολοκληρώσουμε την όλη προσέγγιση, ίσως θα μπορέσουμε καλύτερα να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Καλώς. Θα διαβάσουμε προσεκτικά το έγγραφο που θα δώσετε. Ε, είναι καλό που το ελεκτικό συνέδριο έκανε την παρουσίαση και βλέπουμε αυτή την εξέλιξη σε πολλές χώρες. Το ελεκτικό συνέδριο έχει ελεκτικό ρόλο, έλεγχο συμμόρφωσης, αλλά και έχει και άλλες αποστολές, των συμβουλών, παραδείγματο χάρη, συμβουλευτικό ρόλο για τι αποφάσει που λαμβάνονται και εφαρμόζονται και πώ εφαρμόζονται. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ματέ, σα ευχαριστώ και του δύο σα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ε, μονίμως παρακολουθούμε αυτό το θέμα, το θέμα τη οδηγία των υπηρεσιών. Σα ευχαριστούμε για αυτά που μα είπατε. Έχουμε ακόμη ένα σημείο σημαντικό στην ημερήσια διάταξη. Αφορά την προσβασιμότητα. Σύγκληση των νομοθετικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι απαιτήσει προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Ο υποφαινόμενος είναι εισηγητής για το κείμενο αυτό. Και σήμερα θα αφιερώσουμε την ε, συνεδρίασή μας στην ε, αξιολόγηση της μελέτης επιπτώσεων, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων. Και μάλιστα έγινε μια προκατακτική συζήτηση για τη μελέτη αυτή και τέθηκαν ερωτήσεις από πολλούς συναδέλφους, ε, προβληματίστηκαν για αυτή τη μελέτη επιπτώσεων ε, για το πώς είναι παροχημένη τη μεθοδολογία που ακολούθησε και ούτω, καθε, καθεξής. Οι εσωτερικές υπηρεσίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η υπηρεσία EPRS ε, έκανε μία μελέτη επί της μελέτης επιπτώσεων και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο για να μας την παρουσιάσει. Από μακριά δυστυχώς δεν βλέπω το όνομά σας. Κυρία Μανιάκη. Δύο έχετε έρθει. Παρακαλώ, περιμένουμε την έκθεση που καταρτήσατε επί της εκθέσεως ε, με επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να κάνουμε την, τον πρώτο απολογισμό της μελέτης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση ε, για την προσβασιμότητα. Πριν σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της έκθεσης, θα ήθελα να σας πω ότι ο προκατακτική αξιολόγηση της μελέτης επιπτώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η εκτίμηση της ποιότητας με βάση τους κανόνες που προβλέπονται Στι κατευθυντήρες γραμμέ ε, καλύτερη ομοθεσία για τέτοιε μελέτε επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η εκτίμηση, η αξιολόγηση δεν αφορά την ουσία ή τι επιλογέ πολιτική ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά μόνο την ποιότητα. Εμεί ε, θέλουμε με την δική μα έκθεση να βοηθήσουμε τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, να καταστήσουν μια αντικειμενική ανάλυση για να δουν κατά πόσο οι πληροφορίε και η ενημέρωση τη μελέτη επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έγκυρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κοινοβουλευτική εκτίμηση αυτής της πρότασης. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων για την Ευρωπαϊκή Πρόταση για την Προσβασιμότητα, ε, τα βασικά σημεία της δικής μας αξιολόγησης παρακολουθούν τη δομή της μελέτης επιπτώσεων και επικεντρώνονται σε πέντε συγκεκριμένα σημεία. Καταρχήν, ε, ο λόγος της μελέτης επιπτώσεων και η αιτιολόγηση της πρότασης ε, είναι γενικός καλός, ε, είναι σχολαστική έκθεση, ε, κάνει διάγνωση του προβλήματος που χρήζει κοινοτική αντιμετώπισης, ε, εξαιτήσει του κατακαιρματισμού που υπάρχει για τους κανόνες προσβασιμότητας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, καθώς και για τις δημόσιες προσβάσεις, δημόσιες συμβάσεις στην εσωτερική αγορά. Και μάλιστα ο κατακαιρματισμός θα ε, αυξηθεί μετά τη σύμβαση του ΟΗΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των αναπήρων και ε, περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και στο διατακτικό και στο παράρτημα για τις ε, ισχύοντα και μελλοντικά παραδείγματα κατακαρματισμού για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από την πρωτοβουλία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών εξηγούνται με σαφήνεια και διαφάνεια στο βασικό τμήμα και της μελέτης επιπτώσεων και του αντίστοιχου παραρτήματος. Η μελέτη επιπτώσεων ε, ε, ε, εξηγεί τα τεκμήρια που χρησιμοποίησε για το κόστος των, υπηρεσιών, των επιχει... για τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή του των κανόνων προσβασιμότητα και το κόστο του κατακαιρματισμού. Είναι θετικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να είναι όσο πιο περιεκτική και σχολαστική γίνεται, αλλά η υπερβολική σχολαστικότητα και η πληθώρα των παραδειγμάτων επηρεάζουν κατά τη γνώμη μας την ενάργεια της και τη σαφήνεια αυτής της έκθεσης ε, επιπτώσεων που είναι αρκετά μακροσκελής και μερικές φορές ε, επαναληπτική. 350 σελίδες είναι η έκταση αυτής της ε, και δεν είναι εύκολο να βρει κανεί πληροφορίε ή να τι αντιληφθεί. Η μεθοδολογία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προβλέψει το πώ ε, κράτη χρησιμοποίησαν διαφορετικά στοιχεία προσβασιμότητα για προϊόντα και υπηρεσίε ε, και θα το κάνουμε μέχρι το 2020, δεν είναι η πληροφορία σε αυτές και πρέπει να γίνει πολύ αναλυτική μελέτη για να καταλάβει κανεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα καλύπτει μόνο μερικές υπηρεσίε. Ε, Πιστεύουμε ότι αν είχε αναλυθεί καλύτερο αντίκτυπος ε, του ισχύοντος κατακαιρματισμού και, τη, και της ε, συνέπειας ε, στην λειτουργία της αγοράς ήταν πιο αποτελεσματικός για να έχουμε καλύτερη αντίληψη του πόσες επιχειρήσεις επηρεάζονται. Βέβαια ο σύνδεσμος μεταξύ του κατακαιρματισμού και της εφαρμογής της σύμβασης του ΟΗΕ θα έπρεπε να είναι πιο αναλυτικός. Αυτό το αναφέρει και το Συμβούλιο Μελέτη Επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη θετική γνωμοδότηση που έδωσε επί τη έκθεση τον Ιούλιο του 2013. Γενικώ πάντω η έκθεση είναι μεστή και συνάδει με του βασικού τους βασικούς στόχους που είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση ε, της πρόσβασης ε, των αναπήρων. Και μάλιστα η αιτιολόγηση της ε, κοινοτικής παρέμβασης και η προσθέμενη αξία τη κοινοτικής παρέμβαση αναλύονται επαρκώς, καθώς και τα θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας. Όλα αυτά ε, αναλύονται δεόντως στα αντίστοιχα τμήματα. Η αναλογικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μελέτη επιπτώσεων κατά την υιοθέτηση κάποιων επιλογών πολιτικής. Και επίσης ε, προτείνονται διασφαλιστικές δικλείδες για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μην ε, υποστούν τι αρνητικέ συνέπειε υπερβολική επιβάρυνση από την εφαρμογή αυτή τη πρωτοβουλία. Βέβαια, η μελέτη επιπτώσεων θα μπορούσε να είναι πιο αναλυτική ω προ το πώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, μπορούν ε, να, παρουσιάσουν αυτή τη δυσανάλογη εφαρμογή στην πράξη. Σε ό,τι αφορά τι επιλογέ πολιτική. Οι συγκεκριμένε επιλογέ πολιτική ε, συνάδουν με τον ορισμό του προβλήματο και μαζί με την επιλογή της μη περαιτέρω εξετάστηκαν ε, οι μη κανονιστικές ε, προτάσεις, συστάσεις, καθώς και κανονιστικές, ε, δηλαδή οδηγίες ή είτε οδηγίες έμεσης είτε άμεσης εφαρμογής για τη ρύθμιση της προσβασιμότητας. Είναι σαφές από την αρχή του κειμένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά την οδηγία από τις άλλες επιλογές πολιτικής αλλά δεν ε, προτιμά ένα από τα δύο ίδια οδηγιών. Κάνει μια σύγκριση μεταξύ των στοιχείων των δύο διαφορετικών επιλογών και αναφέρεται υπέρ και τα κατά. Βέβαια, οι επιλογές αυτές είναι σαφείς, αλλά ίσως θα μπορούσαν να είναι πιο αναλυτικές πληροφορίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελέτη επιπτώσεων για το πώς η προτινόμενη χρήση του ε, σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα των Ευρωπα... στα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να μην μπερδεύονται οι καταναλωτές ότι αφορά διαφορετικές χρήσεις του σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων, η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως οικονομικά στοιχεία, ίσως εις βάρος μιας πιο ευρυθούς ανάλυσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αντικτύπων. Βέβαια αυτό θα ήταν αναμενόμενο μάλλον, μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρότασή της επικεντρώνεται στο θέμα της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να ποσοτικοποιήσει τα πράγματα και υπολόγισε τις οικονομίες από κάθε επιλογή πολιτική σε σχέση με το βασικό σενάριο. Επίσης, ε, ε, εκτίμησε το κόστος ε, για τις επιχειρήσεις για να δώσουν πληροφορίες προσβασιμότητας, αναπροϊόν η υπηρεσία με βάση τις διάφορες επιλογές πολιτικής, εκτιμώντας το κόστος αυτό 18 ευρώ την ώρα. Μία βέβαια μεγαλύτερη μεθοδολογική ανάλυση για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των 144 ε, και το 1.400 ευρώ διοικητικό άχθος ε, ανά επιχείρηση για κάθε μία από τις διαφορετικές επιλογές θα ήταν ευπρόσδεκτη. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη επιπτώσεων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο των ε, επιλογών αυτών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έγινε μια δημοσκόπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα θέματα αυτά, αλλά δεν φαίνεται ότι κατέληξε σε ποσοτικοποιημένη ανάλυση του κόστους ωφέλους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, η οικονομική ανάλυση αυτή καθ' αυτή επικεντρώνεται περισσότερο στις οικονομίες, στην εξοικονόμηση που γίνεται. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να διαρευνηθεί και το κόστος για τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη της πρότασης. Ιδιαίτερα όταν έχουν ε, ήδη ρυθμίσει το θέμα αυτό της προσβασιμότητας και τι θα ε, συνεπάγεται η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες προσβασιμότητας. Αυτό το επισήμανε και το Δαντιστικό Συμβούλιο ε, Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν την ανάλυση και οι διάφορες επιμέρους μελέτες είναι σχετικά παροχημένα. Οι περισσότερες μελέτες, μάλιστα, είχαν γίνει πριν από το 2010. Και μάλιστα η έκθεση Deloitte στηρίζεται σε δεδομένα της αγοράς του 2011 και αναφέρεται γενικώ και το πανεπιστημιακό δίκτυο για τα άτομα με αναπηρίες. Αλλά τα στοιχεία αυτά αναγόνται και αυτά στο παρελθόν, στο 2012. Οπότε θα ήταν χρήσιμο αν έγινε κάποια επικαιροποίηση των στοιχείων των προηγούμενων μελετών. Γιατί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ε, τις πρωτοβουλίες αφορούν ε, την ψηφιακή εποχή, ενώ οι εκθέσει είναι πιο παροχημένες. Σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, ε, η μελέτη επιπτώσεων ε, αποδεικνύει εκτενείς διαβουλεύσεις, ανοιχτές και δημόσιες, που κράτησαν 8 εβδομάδες, που έγιναν το 2011 και αρχές του 2012, με επιτυχία έκβαση. 821 απαντήσεις δόθηκαν Επίση, ε, έγιναν και συναντήσεις υψηλού επίπεδου με εκτελεστικού διευθυντέ ε, επιχειρήσεων και μια δημοσκόπηση και από το Ευρωβαρόμετρο. Μάλιστα με 25.000 ε, τηλεφωνικές συνομιλίες στα πλαίσια της έρευνας. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων παρουσιάζονται καλά στην έκθεση, αν και δεν γίνεται κατηγοριοποίηση αυτών. Για παράδειγμα, ε, θα μπορούσαν να ληφθούν καλύτερη υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Πάντως, ο τελικός κατάλογος προτεραιοτήτων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προτεραιότητες και των ενδιαφερομένων, όπως ε, προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά τη συνοχή μεταξύ της μελέτης επιπτώσεων και της νομοθετικής πρότασης, φαίνεται ότι η νομοθετική πρόταση συνάδει με τη μελέτη επιπτώσεων και σε μεγάλο βαθμό ε, ακολουθεί τις συστάσεις της μελέτης επιπτώσεων. Και μάλιστα η οδηγία είναι η δράση που επιλέχθηκε σε ό,τι αφορά τώρα τι υπηρεσίε φιλοξενία που περιλαμβάνονται στον τελευταίο κατάλογο προϊόντων και αγαθών ε, και υπηρεσιών τη μελέτη επιπτώσεων, ε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην κυρίω πρόταση. Και επίση υπάρχει ένα προαιρετικό στοιχείο για τα κράτη-μέλη στην πρόταση, ενώ στη μελέτη επιπτώσεων προέκυπτο δεσμευτικό. Η μελέτη επιπτώσεων έλεγε ότι ε, τα κράτη-μέλη όφυλαν να το καλύψουν το περιβάλλον προσβασιμότητας τα προτερήματα της μελέτης επιπτώσεων. Η επιθυμία διαφάνειας, οι ευρείες διαβουλεύσεις, η γενική συνάφεια μεταξύ της ορισμού του προβλήματος, η αιτιολόγηση της παρέμβασης, οι στόχοι και οι επιλογές που εξετάστηκαν. Τώρα κάποια στοιχεία που ίσως θα μπορούσαν να ανηλυθούν περαιτέρω ή πιο σχολαστικά σε σχέση με τις παροχημένες εκθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν, την οικονομική ανάλυση που επικεντρώνεται κυρίως στην εξοικονόμηση, το σύνδεσμο μεταξύ του κατακαιρματισμού και της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και ίσως κάποιες πιο ενδελεχείς πληροφορίες για το πώς το σήμα ε, και ε, το θέμα της, αναλογικ... της, ε, αυτο... της ε, εκτίμησης αναλογικότητας από τις ίδιες επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτά και είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειαστείτε στο μέλλον είτε περαιτέρω μελέτη επιπτώσεων είτε πιο σχολαστική αξιολόγηση της μελέτης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων ή μελέτη επιπτώσεων συγκεκριμένων ε, τροπολογιών της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας κάνουμε να δουλέψετε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που μου το προτείνετε ίδια. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιδράσει στην παρέμβασή σας. Και μετά θα θέσω κάποιες ερωτήσεις και στους συναδέλφους. Alors, euh, je vais passer la parole à Madame euh, Emmanuelle Grange, qui euh, représente la Commission. Ε, Grange, που εκπροσωπεί ε, Merci, c'est Manuela Gilling. Manuela ε, Gilling. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν προφέρα στα το όνομά σας. Θα μιλήσω αγγλικά. This, ε, ε, Ευχαριστώ για την συνοπτική παρουσίαση της αξιολογήσεως που Θα επανέλθω σε κάποια στοιχεία που αναφέρατε να εξηγήσω περαιτέρω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφερθήκατε στη χρήση του σήματος Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την προσβασιμότητα, για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές. Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, CE, δείχνει συμμόρφωση με κάποιους προκαθοριστέντες κανόνες. Άρα, η ενημέρωση των καταναλωτών και οι πληροφορίες που διατίθενται δεν διατίθεται μέσω του σήματος CE, αλλά συμπεριλαμβάνονται στις προϋποθέσεις προσβασιμότητας και στους όρους και απαιτήσει προσβασιμότητας. Για το κόστος, κάτι σημαντικό. Οικονομίες και κόστος, εξοικονομήσεις ποσών και κόστος και πώς συνδέεται με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ανέλαβαν υποχρεώσεις. Αυτό συνεπάγεται ένα κόστος. Τι λέει η Σύμβαση? Ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την προσβασιμότητα. Αυτό συνεπάγεται κόστος. Αυτό το νομοθέτημα τι επιτρέπει? Οικονομίες. καθορίζοντας απαιτήσει περί προσβασιμότητας που θα ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι διευκολύνεται το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών και αγαθών. Γι' αυτό γίνεται λόγος για οικονομίες και όχι κόστος. Για δυσανάλογο βάρος το δυσανάλογο αυτό άχθος αναφέρεται στην ίδια την πράξη πώς αντιμετωπίζεται. Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα δυσαναλόγου βάρους. Γιατί είναι στην αξιολόγηση συνεπιών η στέγαση και όχι στην πρόταση και σχετικές, παρουσίες, σχετικές υπηρεσίες. Όταν εξετάσαμε θέμα της αναλογικότητας και θεωρήσαμε ότι δύο αυτές πτυχές δεν συμπεριλαμβανόταν. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν κατά πόσο θέλουν να έχουν αυτό το περιβάλλον εντός των προβλέψεων ή όχι. Και ε, υπηρεσίες φιλοξενίας δεν συμπεριλήφθησαν διότι θεωρήσαν ότι περισσότερο οι μικρομεσαίες θα συμμετείχαν σε αυτό το τομέα της φιλοξενίας και της στέγασης και αυτό θα ήταν κάτι που θα ήταν δαπανηρό για αυτές. Η εξολόγηση αντιχτύπου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει ένα προς ένα τα διάφορα σημεία του νομοθετήματος. Εδώ κινηθήκαμε ευρύτερα από αυτό που προβλεπόταν στην νομοθετική πρόταση. Uh, Για τα απειρχαιωμένα στοιχεία χρησιμοποίησαμε τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας Όπως ανέφερε και συνάδελφος του Κοινοβουλίου, έγιναν πολλές διαβουλεύσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις. Έγιναν αρκετές συναντήσεις με διάφορους φορείς. Θέλαμε να έχουμε πιο επίκαιρη εικόνα. Όσον αφορά το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών, αν δείτε τη διατύπωση των ορισμών, η διατύπωση είναι αρκετά προσεκτική. Επιτρέπει να λάβουμε υπόψη και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Έχουμε συμπεριλάβει σωστές έννοιες και ορισμούς που καλύπτουν προϊόντα και επιτρέπουν και την χρονική εξέλιξη των προϊόντων, χωρίς να ξεπερνούνται χρονικά οι ορισμοί, να ξεπερνούνται από τις εξελίξεις. Νομίζω ότι απάντησα σε κάποιες από τις εκφραστήσεις ανησυχίες. Θα σταματήσω εδώ και ευχαρίστω να επανέλθω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις προς απάντηση. Καλώς λέει ευχαριστώ πολύ. Είμαι εισηγητής, θα θέσω ερώτηση στο τέλος. Στην κυρία Σενάλοβα θα δώσω το λόγο, που είναι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα των σοσιαλιστών. Eh, eh, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και για τις δύο παρουσιάσεις που ακούσαμε και όντως σήμερα την που δεν αποτελεί την συνήθινη διαδικασία. τη συνήθεια διαδικασία που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ στην Επιτροπή, αλλά θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι ε, τίθενται διάφορα ζητήματα, διάφορα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την πρώτη συζήτηση για τη μορφή που Χαίρομαι λοιπόν που λάβαμε τι πληροφορίε αυτέ και συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι σε κάποιε περιπτώσει δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε μια μελέτη αντικτύπου όπως καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα τα όσα ακούσαμε στην παρούσα φάση θεωρώ ότι ήταν χρήσιμα και ωφέλιμα αφετέρου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε τα πάντα και να εκφράσουμε τα πάντα με αριθμητικά στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταβάλλει φιλετούμε προσπάθειες και είναι άλλωστε και η δουλειά τη. Πιστεύω λοιπόν, όπω ακούσαμε, ότι η μελέτη αντικτύπου προφανώ εστιάζεται στι οικονομικέ πτυχέ και όχι τόσο στον κοινωνικό αντίκτυπο, που πιστεύω ότι είναι και ο πλέον σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή. Μιλάω ε, εκ μέρου των σοσιαλιστών και δημοκρατών στην παρούσα φάση και πρέπει να σας πω ότι προτιμούμε την συνολική προσέγγιση της ε, ενιαίας αγοράς. Υποστηρίζουμε την ε, επέκταση, την εμβάθυνση τη ενιαίας αγορά, αλλά εκ παραλίλου θα πρέπει να τεθούν και οι σχετικές προδιαγραφές ό,τι αφορά τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Υπηρεσίες οι οποίες δεν διατίθενται για όλους τους πολίτες. Στην σύνοψή σας αναφέρεται δικαίω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο το οποίο στο παρελθόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία φιλόδοξη προσέγγιση, μια φιλόδοξη στρατηγική και ότι σε αυτή συγκαταλέγονταν και όλα τα στοιχεία προσβασιμότητα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τα αγαθά για όλα τα κράτη-μέλη. Σημαντικό επίσης είναι να, βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ανέλθουν στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά και τις ε, προδιαγραφές που ορίζονται από τις εθνές συμβάσεις για τους αναπήρους. Ε, άκουσα επίσης στο σχόλιο ότι η μελέτη δικτύπου δεν καλύπτει, δεν συμπεριλαμβάνει και τις απόψεις των αναπήρων των ατόμων τα οποία αφορά ουσιαστικά η μελέτη αντικτύπου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε και εκπροσώπους των ενώσεων, των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους αναπήρους της μελλοντικής μας εργασίας. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπήρειας εκπροσωπεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 18 εκατομμυρίων Ευρωπαίων συμπεριληφθήκε. Ακούστηκε η φωνή του. Έχουμε και την κυβερνητική ομάδα για θέματα αναπηρίας. Τέλος, έγινε μία μεγάλη συζήτηση σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την προκειμένη περίσταση για να ξεκινήσει μια σχετική συζήτηση και ως εισηγήτρια από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Είμαι δεδεθειμένη να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή προκειμένου τελικά να καταλήξουμε στην έγκριση μιας νομοθεσίας που θα επιτρέψει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά με ίσους όρους και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία με τους αγαπητού σκιώδε. Δεν είναι εδώ πέρα ο σκιώδη ε, του ΕΛΚ, αλλά θα πάρει το λόγο ο Αντρέα Σουάμπ από το ΕΛΚ. Λυπάμαι που δεν μπορεί να είναι εδώ ε, ο εισηγητή μα, αλλά διοργανώθηκε τελευταία στιγμή ε, μια συνάντηση των σκιωδών στην οποία έπρεπε να συμμετέχει. Τρεις ερωτήσεις μου ζήτησε η συγκεντρία να θέσω, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι τονίζει στην ε, παροχημένη κατάσταση στην οποία βασίστηκε η μελέτη αντικτύπου, γιατί πρόκειται για στοιχεία από τα έτη 2011 και 2012. Η συνάδελφος Φραήν, λοιπόν, θα ήθελε να γίνει μια επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων πρώτα και να υπάρχουν, λοιπόν, έτσι ενημερωμένα στοιχεία. Κατά δεύτερον, η συνάδελφος Φερχάιν θα ήθελε να γίνει μια οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια αλλαγή και προσαρμογή ασφαλώ έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. και γι' αυτό λοιπόν η κυρία Σαμπίνε Νευραήν θα ήταν λεφτή υπόψη αυτός ο παράγοντας. Και τέλος, η συνάδελφο δεν είναι βέβαιη κατά πόσον ε, η επισήμαση CE αποτελεί τη σωστή λύση και μήπως θα μπορούσε να προκληθεί σύγχυση στους πολίτες γιατί το ΣΥ ουσιαστικά ε, είναι σήμα για την ασφάλεια, όχι για την έλλειψη φραγμών. Αυτές λοιπόν είναι όλες οι βασικές ε, παρατηρήσεις της ε, συναδέλφου και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις περαιτέρω εξελίξεις με μεγάλη προθεμία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Η Κάθριν Στάιλερ. Σας ευχαριστώ. και τον Πρόεδρο και τους προλαλήσαντες. Μία υπενθύμηση. Καταρχήν, τι λέει η σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Στόχος της σύμβασης είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να εξασφαλίσει ίση άσκηση και απόλαυση των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες και με σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας. Άνθρωποι με αναπηρίες, ε, ή με προβλήματα σωματικής ή διανοητικής φύσης δεν θα πρέπει να εμποδίζονται στην πλήρη και αποτελεσματική του συμμετοχή στην κοινωνία ισότιμα με τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους. Αυτό είναι ο στόχος μας σήμερα. Και όταν ακούω και είναι δύσκολο για αυτούς που εξετάζουν περισσότερο τις οικονομικές πτυχές, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφος. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τις κοινωνικέ πτυχέ. και ποιο είναι το κόστος ε, του να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Όταν 14% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει κάποια μορφή αναπηρίας, 45 ε, εκατομμύρια δηλαδή συνάνθρωποι μα έχουν κάποιο ε, είδου αναπηρία. Οφείλουμε να κάνουμε κάτι ώστε όλοι οι συμπολίτε μα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε και αγαθά που για μα είναι δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, τι λένε τα δεδομένα. Υπάρχουν ε, όμως άλλα δεδομένα, γιατί εγώ δεν τα βρίσκω από αυτά που μας ε, έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλουμε επίκαιρες βάσεις δεδομένων, επίκαιρα στοιχεία, ενημερωμένα. Το θέμα των ε, δεδομένων λοιπόν δεν μας θέτει σωστά τις βασικές αρχές της συζήτησης. Θα πρέπει να έχουμε σωστά δεδομένα και να δράσουμε ανάλογα. Σε ό,τι αφορά την τη συμπερίληψη, την αποφυγή του αποκλεισμού, ποιο είναι το κόστος να μην κάνουμε τίποτα. Ποιο θα είναι το κόστος για αυτού του 45 εκατομμύρια συνανθρώπου μας. Γιατί έχουμε τη διακομματική ομάδα για το θέμα αυτό της κινητικότητας και των ανθρώπων με αναπηρία. Θέλουμε λοιπόν εκπρόσωποι ε, των αναπήρων να έρθουν και να μας μιλήσουν για να δούμε και τη δική τους σκοπιά. Και σε ό,τι αφορά τα, τον ψηφιακό κόσμο. Μιλήσατε και για το θέμα των ιστοσελίδων και των ιστοτόπων. Πολλές εφαρμογές αναφέρθηκαν. Κάθε 8 λεπτά, ε, από κάθε 8 λεπτά που ξοδεύει κανείς στο Ιντερνετ, 7 τα αφιερώνει σε μία εφαρμογή. Η οικονομία των εφαρμογών αυξάνεται κατά 24% ετησίως. Οπότε θα πρέπει και οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες να μην αποκλείονται από την πρόσβαση στις ε, εφαρμογές. Γιατί όλο και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται μέσω εφαρμογών και πληροφορίες επίσης δημόσιες. Είδαμε πόσο σημαντικές είναι οι εφαρμογές. Δεν θέλουμε να αποκλείονται 45 εκατομμύρια των συμπολιτών μας επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές. Γιατί είναι σημαντική αυτή η πρόσβαση, θεμελιώδες δικαίωμα και ελευθερία. Τεράστιο το δυναμικό λοιπόν αυτή τη νομοθετική πρόταση, αρκεί να μπει σε σωστέ βάσεις και να επανέλθουμε στο ζητούμενο, στα, στο βασικό μέλημά μα, που είναι η ισότιμη μεταχείριση των ανθρώπων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Κάθριν. Έχω και κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα ε, κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο που είναι η μελέτη επιπτώσεων, η μελέτη αντικτύπου και η μελέτη αντικτύπου επί τη μελέτη αντικτύπου. Η δική μα μελέτη αντικτύπου επί τη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μιλούμε για την ουσία τη νομοθετική πρόταση, αλλά για την ίδια τη μελέτη αντικτύπου. Και η υπηρεσία ερευνών και οι συνάδελφοι έθεσαν εύστοχες παρατηρήσεις ε, για το τι θα πρέπει να μας προβληματίσει σχέση με αυτή τη μελέτη αντικτύπου. και θα χρησιμοποιήσω αυτά τα σχόλια και θα τα παρουσιάσω κάπως διαφορετικά γιατί ως συγητής θεωρώ μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να λάβει υπόψη τη δική μας ε, εκτίμηση της μελέτης αντικτύπου ε, και να επηρεάσει έτσι την νομοθετική της πρόταση. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Οπότε και οι υπηρεσίε φιλοξενίας, παροχής ε, διατροφής που δεν εμπιπτούν ε, ούτε στην οδηγία ή στη μελέτη επιπτώσεων. Να δούμε ίσως το, το θέμα του πεδίου εφαρμογή και πάλι. Αυτό που μας ε, λυπεί είναι ότι ανταλαμβανόμαστε την αρχή της αναλογικότητας, αλλά δεν βλέπουμε εμπράκτος να εφαρμόζεται στους τομείς που αφαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογή. Γιατί αφαιρέσαμε κάποιες υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογή γιατί για αυτούς η αρχή της αναλογικότητας θα καθιστούσε πολύ επιβαρυντική την συμπερίληψη. Αλλά νομίζουμε ότι ήταν κάπως αυθαίρετη αυτή η επιλογή εξαίρεση μερικών υπηρεσιών. Και μάλιστα ήταν κάπως εκ των υστέρων αυτή η αφαίρεση και η επιλογή. Σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις, τις ευρείες διαβουλεύσεις με εκπροσώπους κοινωνία των πολιτών, αλλά και τη δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν ε, αναφέρεται συγκεκριμένα η, γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών ε, που έχουν αναπηρίες. Πώς ένας ανάπηρος πολίτης ε, δίνει τη γνώμη του στις ερωτήσεις που θέτει το Ευρωβαρόμετρο. Πώς γίνεται η ιεράρχηση των τομέων για τους οποίους ε, απαιτείται τέλεια προσβασιμότητα. Γιατί θα πρέπει οι ίδιοι πολίτες που έχουν κάποια αναπηρία να κάνουν αυτή την ιεράρχηση των τομέων στους οποίους ε, χρειάζονται κατεπηγόντως και πλήρη πρόσβαση ή προσβασιμότητα. Γιατί και η γνώμη των αναπήρων θα πληροληφθεί υπόψη είτε μέσω των ε, οργανώσεών τους είτε μέσω μεμονωμένων προσωπικών προτάσεων. Αλλά δεν θέλετε αυτό με σαφήνεια στην μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης και της επιλογής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πειράστηκαν από τη γνώμη των αναπήρων που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι γιατί αυτοί υποφέρουν από την αναπηρία και την έλλειψη προσβασιμότητας εξαιτία της. Και μάλιστα όσοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σήμερα ε, δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που θα είναι αύριο ενδιαφερόμενοι. Γιατί όλοι είμαστε δυνάμοι άτομα με ανάπηρες. Και να πάει στιγμή μπορεί κανείς ε, να μείνει ανάπηρος. Είτε για λόγους σωματικούς είτε για λόγους πνευματικούς. Και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαντικό θέμα και για την Επιτροπή αλλά και για το στόχο της νομοθετικής πρότασης που είναι να δημιουργηθεί μια αγορά για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επεκταθούν στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο να είναι περιορισμένα στην εθνική τους αγορά. Να εντείνουμε τον ανταγωνισμό, τον υγιή ανταγωνισμό για να υποφελθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και καλό θα ήταν υπήρχε και στη μελέτη αντικτύπου μια ανάλυση κόστους κόστος-οφέλους ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι και στο μελλοντικό έργο για την οδηγία, αλλά και στις συναντήσεις που θα έχουμε, και δίκιο έχετε ότι θα πρέπει να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε με τους οικονομικούς τελεστές και φορείς, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μάλιστα μερικές φορές να σταθούμε και στο πλευρό τους πιο δραστήρια και ενεργά. Γιατί ε, είναι περιορισμένες πολλές φορές σε τοπικές εθνικές αγορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να, να προχωρήσουν, να το κάνουν χάρη στην οδηγία, αλλά και εκείνες που δεν το επιθυμούν να βρουν και εκείνες κάποιες διεξόδους. Επίσης, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του σήματος ΕΕ. ΣΥΗ. Αναφερθήκατε μερικέ από το σήμα το ευρωπαϊκό. Α, δεν νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό το σήμα από τον καταναλωτή, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές έννοιες για το σήμα αυτό. Για τους περισσότερους καταναλωτές, το σήμα ε, ε σημαίνει ότι έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι, συνάδει, συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σημαίνει απλώς κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Ενώ στην ουσία το σήμα ε, ε σημαίνει ε, ότι ότι συμμορφώνεται με, τους, ε, με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οπότε θέλουμε το τρίτο σήμα που να λέει συμμορφώνεται με τις απαιτήσει προσβασιμότητας. Δεν ξέρω αν θέλουμε μια τέτοια επέκταση. Θα πρέπει να αντιληφθούμε την αφησιμία που υπάρχει για τη χρήση αυτού του ευρωπαϊκού σήματος. Γιατί ε, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει ε, τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη χρήση του σήματος αυτού. Ίσως θα το δούμε επευκαιρία του, της εξέτασης νομοθετικής πρότασης. Ίσως θέλουμε ένα, επιπλέον λογότυπο στο σήμα ΕΕ που να δείχνει το ιδιαίτερο μας ενδιαφέρον για τους αναπήρους. Και να έχουμε με το σήμα αυτό όχι μόνο συμμόρφωση ασφάλεια, αλλά μια ευρύτερη συμμόρφωση και με τι απαιτήσει προσβασιμότητα προκειμένου. Αλλά έτσι θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε ή να υπεραπροσδιορίσουμε το σήμα αυτό από την αρχή. Γιατί αν δώσουμε διαφορετικό νόημα για το θέμα της προσβασιμότητας, αυτή, αυτό το διαφορετικό νόημα ίσως μεταφερθεί και σε άλλους τομείς. Και να ολοκληρώσω με ένα σημείο που ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι και που κατά τη γνώμη και το μείζον ζήτημα. Το θέμα της ε, αρχαιότητας αυτών των δεδομένων. Είναι παροχημένες οι εκθέσεις που αποτέλεσαν τη βάση των στοιχείων. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ε, πολύ παρατεταμένη προθεσμία και το, χρόνο, το μεγάλο χρόνο που χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τότε υποσχέθηκε το κείμενο και όταν το ετοίμασε. Γι' αυτό και τα στοιχεία έχουν ξεπεραστεί. Απ' τη μια επικεντρώνουμε τη δράση της νέες τεχνολογίες, ε, και την ψηφιακή εποχή και από την άλλη χρησιμοποιούμε πεπερασμένα στοιχεία, παροχημένα, προτετραετίας. Αν λάβουμε υπόψη τα smartphones, αυτά τα τηλέφωνα που είναι και ένας από τους στόχους της οδηγίας. Με τα τηλέφωνα αυτά, τα smartphone, έχουμε προχωρήσει πολύ σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε συγκεκριμένες λειτουργίες με τα smartphone, σήμερα κάνουμε άλλα πράγματα. Και μια και η οδηγία αυτή θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να δρομολογηθεί και να μεταφερθεί στι εσωτερικέ ένωμε μετά από μερικά χρόνια θα είναι τελείω διαφορετική ακόμη η χρήση των κινητών, των έξυπνων κινητών. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα μείνουμε ακόμη πιο πίσω και θα έχουμε ήδη μια διαφορά μεταξύ των πρωτοτραετίας μελετών και της σημερινής μελέτης επιπτώσεων και άλλες διαφορές μεταξύ σημερινής μελέτης επιπτώσεων και της ε, στιγμής ε, θέσης σε ισχύ της οδηγίας. Οπότε δεν έχουμε μόνο τετραετή υστέρηση, αλλά οκταετή μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία. Θα έχουμε οκταετή διαφορά μεταξύ των μελετών και της εφαρμογής της οδηγίας. Θα είναι ακόμη πιο παροχημένα λοιπόν τα στοιχεία των μελετών. Οπότε ήθελα να ζητήσω από την υπηρεσία ερευνών μας να μας να μας πει και αφού έχει εξετάσει το θέμα, να μας πει είναι δυνατόν να γίνει μια επικαιροποίηση, μια ενημέρωση των στοιχείων και με ποιο τρόπο. Δεν λέω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει η υπηρεσία των ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά ε, διαρωτώ με, είναι δυνατόν και κάπως σύντομα σχετικά να έχουμε μια μεθοδολογία ώστε να μην ε, ήδη από την αρχή έχουμε μια τετραετή στέρηση και διαφορά σε σχέση με τα στοιχεία, γιατί αυτό θα μα ε, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, γιατί στο μέλλον η αρχική καθυστέρηση θα προσθεθεί στην μελλοντική μέχρι τη θέση σε ισχύ του κειμένου. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος ακόμη και θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να λάβει και πάλι το λόγο για να σχολιάσει τις παρατηρήσεις μας πολύ ευχαρίστως. Μάλιστα έκανα και λάθος πριν, γιατί Άλλο όνομα μου είχαν δώσει συνάδελφοι και σας είχα αποκαλέσει με διαφορετικό επώνυμο. Σας ζητώ και πάλι συγγνώμη. Problem, really. Thank you for giving me a second time uh, the floor. Um, just quickly a few points. Σας ευχαριστώ. Λίγα σημεία ήθελα να δείξω. Ένα θέμα και μία ερώτηση τέθησα για τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό αντικτύπο. Αυτό καλύπτεται στη μελέτη αντικτύπου ο κοινωνικός αντικτυπός είναι πολύ θετικός, ε, ο περιβαλλοντικός είναι αμεληταίος. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει με μέση αντικτύπο. Τα άλλα σημεία αφορούν τις κοινωνικές πτυχές, τις οποίες ενδεχομένω να μην τις τονίσαμε επαρκώς, η συνθήκη που θέλει να επιφέρει η συνθήκη του ΟΙΕ. Σκοπός είναι να τεθούν κανόνες που θα προωθήσουν τα προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Και εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι καταναλωτές, τα άτομα που έχουν λειτουργικές αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρίες ή με λειτουργικού περιορισμού, άτομα με αναπηρίες ή οι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από μια ευρύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών από καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές. Άρα, είναι σαφής ο στόχος να βοηθηθούν οι άνθρωποι με αναπηρή ή με λειτουργικούς περιορισμούς. Και αυτό το νομοθετήμα δεν θα είχε προκύψει χωρίς ε, τη σχετική συνθήκη του ΟΗΕ για τα αναπηρά άτομα. Για το θέμα ανάλυση κόστου ωφέλου σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε. Αυτό περιλαμβάνεται στη μελέτη δικτύπου. Παράτημα 2, σελίδα 178. η μελέτη που λαμβάνει υπόψη και το πότε το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στις ρυθμίσεις αυτές και ποιος είναι ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί στις ρυθμίσεις. Για τα δεδομένα τώρα. Όπως είπα και πριν, χρησιμοποίησαμε τα δεδομένα που είχαμε στην διάθεσή μας. Είχαμε πάρα πολύ, πολλές διμερείς επαφές με ενώσεις και οργανώσεις ε, αναπήρων, EDF, ε ε, μη κυβερνητικές high level group για την αναπηρία και τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στη μελέτη αντικτύπου χρησιμοποιούνται για να προβληθεί το ποια θα είναι η κατάσταση το 2020, γιατί βλέπουμε ότι ο κατακαιρματισμός που επικρατεί στην αγορά ε, σίγουρα θα αυξηθεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συνθήκης του ΟΗΕ. Άρα πραγματικά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα σε ό,τι αφορά τον ορισμό και το κατά πόσον οι ορισμοί εξακολουθούν να είναι επίκαιροι και ενημερωμένοι. Να σας πω ότι για τα εφή κινητά τηλέφωνα βλέπουμε ότι αποτελεί τραυματικές συσκευές που συνδέονται με τηλεφωνικές υπηρεσίες. Ε, ακούγεται πάρα πολύ περίπλοκο αυτός ο ορισμός, αλλά ουσιαστικά σκοπό έχει να καλύψει το, τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, όπως, του ευθύου τηλεφώνου, όπως το γνωρίζουμε σήμερα σε δύο χρόνια. Αυτή την προσέγγιση ακολουθούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς θα επανέλθουμε επί του θέματος διότι στο πρόγραμμά μας προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού το Σεπτέμβριο και το σχέδιο εκθέσεως που θα σας υποβάλω θα υποβληθεί αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί το θέμα αυτό και οι συζητήσεις με τις τροπολογίες τέλος Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε συνεχεία στην Ήμικο. Ιδού Ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα. Να συμφωνήσουμε επί του προγράμματος, το γνωρίζετε ήδη. Επόμενη συνεδρίαση 13 Ιουνίου το απόγευμα και 14 Ιουνίου πρωί και απόγευμα εδώ στα συνηθισμένα μας ωράρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.